So, wir haben ein strammes Programm heute. Κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας είναι φορτωμένο λοιπόν σήμερα, ελπίζω και θα ήθελα να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η σημερινή ακρόαση Right to Water μεταδίδεται στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καταρχάς θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους ε, υπεύθυνους της πρωτοβουλίας αυτής και την κυρία Αν-Μαρή Περέτ. Καλώς ορίσατε κυρία Αν-Μαρή Περέτ, καλώς ορίσατε. Θα ήθελα εξ αρχής να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ που μου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα καταφέρατε να συλλέξετε 1,9 εκατομμύρια υπογραφές. Είναι πραγματικά εξαιρετική αυτή η επίδοση για μια τέτοια πρωτοβουλία ιδιωτικής ε, προέλευσης ή οποιασδήποτε προέλευση εδώ που τα λέμε, 1,9 εκατομμύρια υπογραφές. Να καλωσορίσω και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ, ανάμεσά μας, τον κύριο Μάρος Σεφκοβιτς και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κιόλα. Κύριε Σεφκοβιτς, γιατί ήταν ο πρώτος ε, που στην ακρόασή του τότε στην αρχή της θητείας ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο να διευκολύνει κατά το δυνατόν την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία αυτή και να υπάρχει και μια τέτοια δυνατότητα στο διαδίκτυο για την ε, διοργάνωση αυτών. Αυτό το επεξεργαστήκαμε λοιπόν από κοινού εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θεωρώ ότι έχει νόημα να υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αυτής υπογραφής. Στο διαδίκτυο, ιδάλλως, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τέτοιους αριθμούς. Συγκεντρωθήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα για να ακροαστούμε, για να ακούσουμε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Έχουμε εδώ πολλούς συναδέλφους, έχουμε και πολλούς εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε από το δικό μας θεσμικό όργανο. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, η Επιτροπή για το Περιβάλλον, για τη Δημοσιογεία και για τα τρόφιμα συμμετέχουν και η Επιτροπή για την Ενιαία Αγορά και η Επιτροπή ε, Αναφορών. Σήμερα λοιπόν, όπως γνωρίζουμε και από την ακρόαση των Επιτρόπων, θα διαμοιράσουμε λοιπόν τα, το χρόνο μας και θα συζητήσουμε το θέμα του νερού. 1,9 εκατομμύρια υπογραφές έχουν συλλεχθεί έως σήμερα. 1,6 εννέα υπογραφές, ε, εκατομμύρια υπογραφές ε, έχουν κριθεί παραδεκτές. 1,2 εκατομμύρια από τη χώρα μου. Είμαι πολύ περήφανος. Για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό θέμα, ακόμα και στα τοπικά κοινοβούλια ε, που συζητήθηκε το θέμα αυτό, εγκρίθηκαν ψηφίσματα και καθόλου το φάσμα, σε όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων ε, έγινε αποδεκτό το θέμα αυτό. Ούτε ένα κόμμα δεν αντιστάθηκε. Δεν είπε ότι δεν θα συμμετάσχει στην ε, πρωτοβουλία αυτή. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ θετικό μήνυμα και λοιπόν σήμερα στη μέρα αυτή θέλουμε να γράψουμε ιστορία γιατί θα γράψουμε ιστορία γιατί πρόκειται για την άμεση Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και εμείς πώς έχουμε φανταστεί την εξέλιξη τη σημερινή ημέρα να ξεκινήσουμε κατευθείαν την ε, ακρόαση θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πέντε λεπτά. Ύστερα ο Γιώργος Χέφνερ από την Επιτροπή ε, Αναφορών και ύστερα θα μας μιλήσει και ο εκπρόσωπος ε, της πρωτοβουλίας ε, των πολιτών. Θα μας μιλήσει μετά η κυρία Αν Μαρή Περέτ, η οποία και θα μας παρουσιάσει την πρωτοβουλία και μετά θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Καταρχάς, σε τρία τμήματα θα διαιρεθεί αυτή η συζήτηση. εγγύηση για το νερό, δεύτερο τμήμα ε, καθολική πρόσβαση στο νερό και τρίτο τμήμα ε, όχι απελευθέρωση των υπηρεσιών υδροδότησης. Και μετά θα έχουμε δύο γύρους ερωταπαντήσεων με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. σα παρακαλώ να τηρήσετε το χρονικό όριο των δύο λεπτών προκειμένου όλοι να πάρουν το λόγο και στη συνέχεια θα γίνει και μια διαδικασία catch the eye όπως τη γνωρίζουμε από την Ολομέλεια, δηλαδή όποιο τραβήξει την προσοχή του Προέδρου θα πάρει το λόγο προκειμένου να θέσουν και άλλα άτομα ε, κατά το δυνατόν περισσότερα. Μία ερώτηση θα δώσω λοιπόν 5 λεπτά το λόγο για τις γενικές παρουσιάσεις και μετά θα απαντηθούν και οι ερωτήσεις ε, ομαδικά. Θα ήθελα να τονίσω τη χαρά μου για το, το γεγονός ότι συμμετέχουν τόσα πολλά άτομα. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και όλες τις, επιτροπές, τις ε, υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διοργάνωση του γεγονότος αυτού εννοείται και την Γενική Διεύθυνση Ίμπολ, την Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος ε, Αναφορών Ενίας Αγοράς και με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας και αυτή να την ευχαριστήσω καθώς και όλες τις υπηρεσίες οι οποίες κατάφεραν να διοργανώσουν με αυτή τη μορφή τη σημερινή ακρόαση. Ανυπομονώ, ανυπομονώ και θα σταματήσω να εκπέμπω για να ακούσω τι έχετε να πείτε. Τι έχετε να μας πείτε. Καταρχάς λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριο Χέφτερ και μετά να ακούσουμε και για την ίδια την πρωτοβουλία. Νομίζω ότι σήμερα μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Και πολύ ασφαλώς θέλουν, ήθελαν live να συμμετέχουν σε αυτή την πρώτη ακρόαση της πρώτης αυτής της μεγάλης ε, πρωτοβουλίας των πολιτών και ανυπομονώ λοιπόν και προσβλέπω στις επόμενες 3,5 ώρες. Γι' αυτό λοιπόν να δώσω και εγώ το καλό παράδειγμα και να μην μακρηγορήσω. Δίνω το λόγο στον κύριο Μάρος Σεύκοβιτς. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αγαπητέ Ματία, Πρώτα απ' όλα να τονίσω πόσο είμαι ικανοποιημένο που έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο. Να σα πω ότι βλέποντα σα από αυτό το ύψο εντυπωσιάζομαι διότι σπανιότατα βλέπει κανεί, μια αίθουσα τόσο γεμάτη με τόσου ανθρώπου που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Θετική ενέργεια λοιπόν και ενθουσιασμό ε, είναι αυτό που αισθάνομαι και αυτό αισθάνομαι και για την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή Διοργάνωσης αυτής της ε, διάσκεψης, της συνάντησης, που μετά από δύο χρόνια από την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή την θέση σε ισχύ αυτής της διαδικασίας, έχουμε την πρώτη επιτυχία με πολύ, με πολύ σοβαρές προϋποθέσεις και απαιτήσει. Ε, εδώ κινητοποιήθηκαν 1,7 εκατομμύρια πολίτες και από μάλιστα 13 κράτη-μέλη. Βρίσκω αυτούς τους αριθμούς εντυπωσιακού και θα ήθελα να πραγματικά να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την προσπάθεια και την επιτυχία τους. Νομίζω από την παρουσία σας εδώ και την στήριξη των πολιτών που έχουμε δει ξεκάθαρα προς την πρωτοβουλία αυτή, Έχουμε πια μια σαφή απόδειξη ότι το εργαλείο αυτό της συμμετοχικής, συμμετοχικής δημοκρατίας ε, λειτουργεί. Οι πολίτες μπορούν πλέον να εκφράσουν την άποψή τους και να επικοινωνήσουν άμεσα με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Να καθορίσουν τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον κατάλογο αυτών των προτεραιοτήτων. Έτσι, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το δικαίωμα στο νερό και τη σχετική πρωτοβουλία σήμερα. Ξέρετε ότι από τον Απρίλιο του 2012 έχει καταγράψει 22 πρωτοβουλίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε ανησυχήσει κάπως, το είχαμε συζητήσει και με τον κύριο Χέφνερ όταν επεξεργαζόμασταν το σχετικό κανονισμό και φοβηθήκαμε ότι θα πρέπει να μην υπάρξει κατάχρηση του δικαιώματος ε, της πρωτοβουλίας των πολιτών, ότι θα πρέπει να επιλεγούν σωστά τα θέματα. Οι ανησυχίες μας τελικά αποδείχτηκαν εσφαλμένες, διότι είδαμε ότι οι πολίτες είχαν συγκεκριμένες προτάσεις για το περιβάλλον, για την εκπαίδευση, τις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα δικαιώματα των πολιτών και ούτω καθεξής. Θέματα που και πρακτικά είναι και αφορούν άμεσα την ουσία της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. Το δικαίωμα στο νερό είναι η σαφώς πρώτη πρωτοβουλία που πληρούσε όλα τα κριτήρια που έχουμε θέσει. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλε δύο πρωτοβουλίε που έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο υπογραφέ ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι. Πάντω θέλουμε να ευχαριστήσουμε ε, τους διοργανωτές όσων ακόμη και εκείνων που δεν έφτασαν το 1 εκατομμύριο, διότι είναι πολύ αυστηρό αυτό το κριτήριο σίγουρα, αλλά κινητοποίησαν πολλού πολίτε. Ξεκίνησε ένα διάλογο πολιτικού περιεχομένου για θέματα τα οποία είναι σημαντικά για του πολίτε. Αυτή η θετική κινητοποίηση από την πλευρά των πολιτών σαφώς ε, προκαλεί την απόκριση της άλλης πλευράς των αντιπροσώπων τους στα εθνικά, το τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωκοινοβούλιο έτσι και η πρωτοβουλία για το δικαίωμα στο νερό. Όπως είπα και το πρωί, έχουμε ξανασυζητήσει κάποιες από τις δυσκολίες που πρέπει να ξεπεράσουν οι διοργανωτές. Προσπαθήσαμε να τις δούμε και με το Ευρωκοινοβούλιο. Κάποιες ήταν πιο αισθητέ καθώς προτιμάζαμε τον κανονισμό και κάποιες από αυτές μας εντυπωσίασαν στην αρχή όπως ε, η δυσκολία να υπάρξει συλλογή των δεδομένων στο διαδίκτυο, να ξεπεράσουμε το όριο του ενός εκατομμυρίου υπογραφών, να υπάρξει εύκολη πρόσβαση και να είναι φιλικό προς το χρήστη το σύστημα. Όταν λοιπόν αναθεωρήσουμε το σύστημα των πρωτοβουλειών το 2015 θα φροντίσουμε να είναι ακόμη φιλικότερες προς το χρήστη οι διαδικασίες που θα ε, χρησιμοποιούνται. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω βεβαιώνοντάς σας όλους και το Ευρωκοινοβούλιο και τους διοργανωτές και όλους τους πολίτες που μας στήριξαν, που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει τη μέγιστη προσοχή προς την πρωτοβουλία αυτή. Όλες οι γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με τους τομείς που αφορά η πρωτοβουλία αυτή και το πρωί ήταν ε, παρούσες, συζήτησαν με τους διοργανωτές σήμερα και τώρα το απόγευμα Έχουμε τρεις υψηλούς εξωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έρθουν για να σας δώσουν τις προκαταρκτικές τους απαντήσεις, να απαντήσουν και σε δικές σας ερωτήσεις και είχαμε το πρωί την ανταλλαγή απόψεων, σήμερα το απόγευμα έχουμε την ακρόαση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δώσουμε την καλύτερη δυνατή απόκριση στις 20 Μαρτίου όπως απαιτεί και ο κανονισμός. Και πάλι λοιπόν να σας συγχαρώ, να σας ευχαριστήσω για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Βλέπουμε μια απτή απόδειξη ότι το εργαλείο αυτό ε, λειτουργεί. Οι πολίτες έχουν πια στα χέρια τους ένα εργαλείο για να έχουν ε, λόγο στο πώς ε, ε, επηρεάζουν τα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σέφνερ, ο οποίος αντικαθιστά την πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών και είναι και εισηγητής υπεύθυνος για το θέμα αυτό. Για τρία λεπτά έχετε το λόγο. you, Ναι, και θα μιλήσω γερμανικά και πάλι, Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω, αγαπητοί ε, παριστάμενοι και πραγματικά και εγώ έχω εντυπωσιαστεί από την ε, ε παρουσία σας. Ακόμα και αυτή η μεγάλη αίθουσα έχει γεμίσει. Είναι πραγματικά ένα ορόσημο αυτό εδώ σήμερα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Γιατί τι ήθιστε οι πολίτες να ακούν και να βλέπουν τι γίνεται στις ε, Βρυξέλλες τι αποφασίζεται για αυτούς. Και αυτοί είναι, οι πολίτες είναι αυτοί τελικά οι οποίοι πρέπει να τα εκτελέσουν αυτά. Σήμερα λοιπόν για μια φορά αλλάζουμε τους ρόλους και ο Ματίας Γκρότ είπε ότι θα περάσουμε στον τρόπο λειτουργίας αυτό, αν θέλετε, που απλά θα προσλαμβάνουμε τα μηνύματα, θα ακούσουμε τι θέλουν να μας πούν οι πολίτες, οι οποίοι μας αποστέλνουν μηνύματα, τι περιμένουν από εμάς τους ευρωβουλευτές για καλύτερη ρύθμιση πολύ βασικών θεμάτων. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ καθοριστικό αυτό βήμα στο μακρύ δρόμο από την, Ευρώπη, από την Ευρώπη των κρατών και των κυβερνήσεων προς την Ευρώπη των πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτής της Ευρωπαϊκής Πρωταβουλίας και να πω ότι πίσω από τα άτομα τα οποία είναι εδώ πέρα σήμερα ε, υπάρχουν άλλα 1,1 εκατομμύρια άτομα τα οποία στηρίζουν τις ελπίδες τους σε εμά για να εισακουστεί η έκκλησή τους και πρόκειται για ένα καθοριστικό ζήτημα το οποίο είναι πάντα και ήταν πάντα σημαντικό και θα είναι πάντα σημαντικό για την ανθρωπότητα. Το νερό είναι λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για τη ζωή. Χωρίς το νερό δεν υπάρχει ζωή και γι' αυτό λοιπόν ε, ανακύπτει όλο και πιο πολύ αυτό το ερώτημα σε ποιον ανήκει το νερό, ποιος ρυθμίζει την πρόσβαση στο νερό και ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι όλοι έχουν την ίση πρόσβαση, ίση πρόσβαση στο νερό. Είναι λοιπόν το νερό ένα ανθρώπινο θεμελιώδες δικαίωμα. Δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί και θα πρέπει να μείνει στα δημόσια χέρια. Λοιπόν, και γι' αυτό σήμερα θα συζητήσουμε σήμερα στα πλαίσια της πρωτοβουλίας. Θα θέσουμε ερωτήσεις θα ακούσουμε, θα μας παρουσιάσει πρωτοβουλία τις δικές σας ε, τοποθετήσεις και πραγματικά ανυπομονώ. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια διοργάνωση μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και σίγουρα όμως θα είναι η τελευταία αυτή η πρωτοβουλία. Αυτή η ακρόαση λαμβάνει χώρα ενώπιον των ειδικών επιτροπών και της Επιτροπής ε, Αναφορών προκειμένου να υπάρχει αδικηματική εμπειρογνωμοσύνη αλλά για να συμμετέχουν να συμμετέχει και η ευρωβουλευτές. Πρωτού ξεκινήσουμε θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν για, την, για τον κανονισμό ECI, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και θα ήθελα κυρίως τους διοργανωτές ε, της πρωτοβουλίας για το δικαίωμα στο νερό αλλά και τους πολίτες, τα σχεδόν δύο εκατομμύρια πολίτες που κρύβονται και απευθύνθηκαν σε εμάς εδώ στο Κοινοβουλίο, να τους ευχαριστήσω λοιπόν και να ελπίζω να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος, κύριε Χέφνερ. Επόμενος ομιλητής, η Αν Μαρή Περέτ, η οποία και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής των Πολιτών και έχει το λόγο για 10 λεπτά για να παρουσιάσει την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Γκρότε. Είμαι πρόεδρος ε, που πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί τα μάλα, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπει κανείς μια κατάμεστη αίθουσα, κάτι που αποδεικνύει ότι έχουμε δίκιο να θέτουμε αυτή την ερώτηση και αυτή την αξίωση, αυτή τη βασική απέτηση για αυτή την πρώτη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών, το δικαίωμα σε πρόσβαση, σε πόσιμο είδωρ και αποχέτευση ως αναπαλωτρίωτα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία τον τρόπο με τον οποίο οργανωθήκαμε γιατί η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ξεκίνησε κυρίως από την δική μας Ομοσπονδία Συνδικάτων των Ευρωπαϊκών Κοινοφελών Υπηρεσιών, αλλά δεν ήμασταν οι μόνοι οργανωτές, δεν ήμασταν οι μόνοι που ξεκινήσαμε αυτό το διάβημα και αυτόν τον αγώνα. Μη κυβερνητικέ οργανώσεις και πολύ σημαντικές μάλιστα μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, όπως η European Antipoverty Network, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καταπολέμησης Φτώχειας, το Ευρωπαϊκό Περιβαλλοντικό Γραφείο, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία και η Ευρώπη για το Κοινό Μέλλον. Είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις που μας συμπαραστάθηκαν στην διοργάνωση αυτή και επίσης και συνδικάτα και η Ευρωπαϊκή Συνομοσποδία Συνδικάτων καθώς και η Διεθνής των Κοινοφελών Υπηρεσιών, η ΕΣΠΕ, μας βοήθησε και μάλιστα η Ρόζα Παρανέλ θα σας μιλήσει σε λίγο ως Γενική Γραμματέας αυτού του φορέα. Φαντάζομαι γνωρίζετε πάνω κάτω τι εστί ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Μας ε, το υπενθύμησαν άλλωστε και οι προλαλήσαντες. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε συγκεντρώσει σχεδόν 1.900.000 υπογραφές και σε λιγότερο από ένα χρόνο, σε 8 μήνες στην ακρίβεια, είχαμε ήδη ξεπεράσει το 1.000.000 εκατομμύριο υπογραφές. Όντως, είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Και αν σκεφτείτε βέβαια πώς οι πολίτες κατοικούν στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα εκατομμύριο, σχεδόν δύο εκατομμύρια δεν είναι και μεγάλος αριθμός. Αλλά ήταν η πρώτη πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών. Και το να καταφέρει κανείς να κινητοποιήσει 2 εκατομμύρια ανθρώπους, σας διαβεβαιώ ότι δεν είναι αμεληταία προσπάθεια και πραγματικά εν τη ισχύς και γι' αυτό ε, χρειαστήκαμε πολύ σημαντικούς συμμάχους ε, στην προσπάθεια αυτή και στάθηκαν στο πλευρό, μας, στο πλευρό μας όχι μόνο τα συνδικάτα αλλά και η κοινωνία των πολιτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και πραγματικά χαιρόμαστε για αυτή την υποστήριξη. Όταν ε, εγκαινιάζεται μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών γίνεται και συγκεκριμένο στόχο. Είναι για να συμπεριληφθεί ένα, πρόγραμμα στο, ένα θέμα στο πολιτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποβληθεί στη συνέχεια μια νομοθετική πρόταση. Και αυτό ξεκινήσαμε να συζητούμε σήμερα ήδη από το πρωί με τον Επίτροπο Σεύτσοβιτ, στα πλαίσια μιας ανταλλαγή απόψεων που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό κάνουμε και τώρα σήμερα σε αυτή τη δημόσια ακρόση χάρη στη διοργάνωση αυτή που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί λοιπόν διαλέξαμε το νερό. Όπως μας υπενθύμισε ο κύριος Χέφνερ, το νερό είναι το απολύτως απαραίτητο στοιχείο, η εκ των όνων προϋπόθεση για οποιαδήποτε μορφή ζωής. Δυστυχώς όμως, εξαιτία των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, το νερό είναι ένας τομέας ε, που απειλείται περισσότερο από ε, πολλούς άλλους. Και δεν μιλούμε μόνο για τις τεχνικές πτυχές της διαχείρισης του ύδατος και της αποχέτευσης, που είναι θέματα δημόσιας υγείας. Το θέμα όμως είναι να εξασφαλίσουμε και πρόσβαση όλων απαρέγκλητα των πολιτών σε πόσιμο είδωρ και σε ένα σύστημα, σωστό σύστημα αποχέτευσης. Και μάλιστα μια στιγμή που η κρίση δυστυχώς συνεχίζεται και συνεχίζει να οξύνει και να εντείνει τις ανισότητες ε, στην Ευρώπη και σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα, το τομέα του νερού. Αυτό που θα ήθελα να κάνω θα ήταν να ξεκινήσω με μια σχετικά γενική παρουσίαση που στη συνέχεια θα την εξειδικεύσουν οι υπόλοιποι ομιλητές μας που θα επικεντρωθούν στα τρία κεφάλαια που ανέφερε ο Πρόεδρος. Θα ήθελα λοιπόν να σας υπενθυμίσω εν συντομία τους λόγους για τους οποίους ε, αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία με 1.659.587 ε, υπογραφές και δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τα 2 εκατομμύρια γιατί έχει κλείσει η προθεσμία για τη συγκέντρωση των υπογραφών. Έχει κλείσει η προθεσμία για τις υπογραφές, αλλά η συζήτηση τώρα ξεκινά στην ουσία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στη συνέχεια θα σας μιλήσω για το τι συνέχεια θα θέλαμε να δώσουμε σε αυτό το διάβημα που είναι πραγματικά ένα διάβημα στα πλαίσια της συμμετοχικής δημοκρατίας. Γιατί στόχος μας είναι να θεσπιστούν δεσμευτικές νομοθετικές διατάξεις για την έμπρεκτη εφαρμογή αυτών των θεμελιδών δικαιωμάτων που είναι η πρόσβαση στο είδωρ, σε πόσιμο είδωρ και στην αποχέτευση το σημείο αφετηρίας της δράσης μας. Στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, Ομοσπονδία μάλλον, Συνδικάτων των Κοινοφελών Υπηρεσιών και σε συνεργασία και συμφωνία με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που σας προανέφερα, εδώ και πολύ καιρό ασχολούμαστε με το θέμα της αναγνώρισης του ύδατος ως αναπαλωτρίο του ανθρώπινου δικαιώματος. Η δυνατότητα αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης Λισαβόνας να οργανωθούν πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών, καθώς και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών του 2010 που αναγνώρισε το είδωρ και την αποχέτευση ως ανθρώπινα δικαιώματα, ήταν και τα σημεία αφετηρίας της δικής μας δράσης. κρίναμε σκόπιμο και απαραίτητο να οργανώσουμε μια πανευρωπαϊκή δράση για να αποκλείσουμε το νερό από την εσωτερική αγορά και να ξεπεράσουμε την οδηγία πλαίσιο για το νερό του 2000 που ήδη αναγνώρισε, όπως αναφερόταν, ότι το νερό δεν είναι ένα συνηθισμένο εμπορικό αγαθό, εμπορεύσιμο αγαθό, αλλά ένα, μια κληρονομιά που θα πρέπει να τύχει προστασίας, προάσπισης και μεταχείρισης ανάλογης. Και μάλιστα στα πλαίσια τη αναθεώρηση τη οδηγία για τι παραχωρήσει, οι επίτροποι Μπαρνί και Ποτότσιγκ μα υπενθύμησαν ότι οι αρμόδιε αρχέ είναι κυρίαρχοι των επιλογών του ό,τι αφορά την παροχή ίδρυυση και οργάνωση ε, των υπηρεσιών του νερού και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν είχε την πρόθεση να επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση του νερού. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η ίδρυυση και η πρόσβαση στην ίδρυυση και την αποχέτευση είναι θεμελιώδεις ε, κοινοφελείς υπηρεσίες. Οπότε θα πρέπει οι δημόσιες αρχές να ασκούν έναν ουσιαστικό έλεγχο στις υπηρεσίες αυτές και επίσης οι πολίτες θα πρέπει να απολαμβάνουν ε, λογικές τιμές που θα αντιστοιχούν στην ικανοποίηση των πρωταρχικών τους αναγκών και όχι στις αποδοχές των μετόχων στα πλαίσια μιας ιδιωτικής διαχείρισης που θα έχει εκχωρηθεί σε μια πολυεθνική εταιρεία. Δυστυχώς ε, πολλοί είναι οι συμπολίτε μας που δεν έχουν πρόσβαση σε ε, πόσιμο είδωρ και σε αποτελεσματικά συστήματα αποχέτευσης. Μπορεί να μην έχουμε ακριβείς στατιστικές, αλλά υπολογίζουμε ότι γύρω στο 1 εκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό και 8 εκατομμύρια δεν ε, απολαμβάνουν ε, ποιοτικό νερό ή ποιοτική ίδρυυση. Δυστυχώς, ε, αν πριτανεύσει η λογική της αγοράς, δεν θα διστάσει κανείς να κόψει το νερό σε οικογένειες που πλήττονται όλο και περισσότερο από τις οικονομικές δυσχέρειες, την αβεβαιότητα και τη φτώχεια. Και μάλιστα η συνέχιση της κρίσης επιδεινώνει αυτές τις ανισότητες και εξασφάλιση τέτοιων κοινοφελών υπηρεσιών γίνεται όλο και πιο προβληματική. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ίδρυυση και η διαχείριση του νερού δεν θα πρέπει να εντάσσονται στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και δεν θα πρέπει να τύχουν απελευθέρωση οι υπηρεσίες του νερού. Αυτά θα είναι τα θέματα που θα αναλύσουν πιο ειδικά οι συνάδελφοι από την Επιτροπή των Πολιτών. Θεωρούμε ότι η παροχή ύδατος και η αποχέτευση δεν θα πρέπει να τύχουν απελευθέρωση. Επαναλαμβάνω εν συντομία τις απαιτήσει μας και τις διεκδικήσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρχικά και μετά σε παγκόσμιο επίπεδο. θεσμι... Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε όλοι απαρέγκλητα οι πολίτες της ε, Ένωσης να έχουν πρόσβαση στο είδωρ και στην αποχέτευση. Και όταν μιλάω για νερό εννοώ πόσιμο νερό και μάλιστα ποιοτικό πόσιμο νερό. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπιστεί υποχρεωτική νομοθεσία για την έμπρακτη και ουσιαστική εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο πόσιμο νερό και στην αποχέτευση, όπως προσδιορίσε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο ψήφισμα του Ιουλίου του 2010. Η διάσπαση, η σαλαμοποίηση, ε, ο τεμαχισμός ή ο κατακαιρματισμός που είναι συνήθως μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από την ε, εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ίδρυυση και την αποχέτευση. Το νερό έχει έναν ολοκληρωμένο κύκλο και αυτή η ακαιρεότητα θα πρέπει να διασφαλιστεί. Ο κύκλος του νερού υπήρχε και πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν από την εσωτερική αγορά και πριν ακόμη τη συνθήκη της Ρώμης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτή την πραγματικότητα και να προσαρμόσουμε αντίστοιχα και τις νομοθεσίες μας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε λοιπόν μία προσέγγιση και αυτό νομίζω ότι είναι το στοιχείο κλειδί, το πιο νευραλγικό σημείο της πρωτοβουλίας μας, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση που θα εδράζεται στα δικαιώματα και όχι στην αγορά. Αυτή είναι η εντολή που μας ανέθεσαν οι συμπολίτες μας μέσω αυτής της ε, πρωτοβουλίας ε, Ευρωπαίων πολιτών για το νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα. Επίσης, ε, σε θέματα παροχής και διαχείρισης θα πρέπει αυτή η υπηρεσία να προσφέρει τους πολίτες όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτούς. Η απελευθέρωση θα ευνοούσε περισσότερο τις πολυεθνικές του ιδιωτικού τομέα, εις βάρος όμως των χωριών, των πόλεων ή και των επιτροπών διαχείρισης των υδροφόρων λεκανών και κάτι τέτοιο δεν θα επέτρεπε ένα οικολογικό ή συμμετοχικό πρόγραμμα. Αυτά λοιπόν. Προσπάθησα να συγκεράσω τις δύο παρουσιάσεις μου σε ένα. Θα περάσω τώρα στις διεκδικήσεις μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζοντας αυτό το θεμελιώδες και αναπολωτρίωτο το δικαίωμα της πρόσβασης στο πόσιμο είδωρ και την αποχέτευση θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την αναγνώριση των δημόσιων αγαθών σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτείνει τις προσπάθειές της και να τις ε, επεκτείνει και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου για παγκόσμια και οικουμενική πρόσβαση σε πόσιμο είδωρ και αποχέτευση. Θα πρέπει να προωθηθεί η παγκόσμια συνεργασία με βάση μη κερδοσκοπικές αρχές και με βάση αλληλέγγυα προσέγγιση μεταξύ των παρόχων ε, νερού και των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες, να εφαρμοστούν εταιρικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου ή μεταξύ δημοσίου και δημοσίων φορέων παροχής ύδατος προκειμένου να βελτιώνεται συνεχώς η ποιότητα αυτών των υπηρεσιών. Αυτά κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν εν ολίγης η παρουσίαση της πρωτοβουλια πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών και ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Περέτ. Και μας κάνατε λοιπόν μια κατευθείαν εισαγωγή σε αυτό το θέμα, κυρίως ό,τι αφορά το πρώτο γύρο. Έχουμε λοιπόν τώρα πέντε συναδέλφους, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο με τη σειρά των ομάδων ο κύριος Ζέιμπερ, ο οποίος είναι υπεύθυνος από πλευρά του Κοινοβουλίου για το θέμα του νερού. Σας παρακαλώ τηρήστε το χρονικό όριο των δύο λεπτών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να συγχαρώ εκ βάθους καρδίας ε, τους οργανωτές αυτής της πρώτης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, γιατί αυτό που πετύχατε είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Θα ήθελα ως ε, πρόεδρος της ε, ομάδας για το νερό αυτή στο Κοινοβούλιο να πω ότι ασχολούμαστε με το θέμα του νερού πολύ ε, εντατικά και σε ό,τι αφορά το θέμα της λειτουργικότητας αλλά και σε ό,τι αφορά το θέμα της ποιότητας του νερού. Θα ήθελα κάποιες ερωτήσεις να κάνω. Επιτρέψτε μου όμως να εκφράσω κάποιες σκέψεις. Καταρχάς, θεωρώ ότι αυτό η καθιέρωση του νερού ως αναπαρατρία του θεμελιωδούς δικαιώματος είναι κάτι το οποίο κάθε Ευρωπαίος, κάθε πολίτης του κόσμου αξίζει. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε σε αυτό στο πρωτόκολλο υπαριθμών 9, άρθρο 1 και στο πρωτόκολλο 26 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Έχουμε τονίσει αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά την ε, κανονική τιμή ε, του νερού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι κοινοφελείς σκοποί και υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την διοργάνωση του κλαμπ νερού. Και πρέπει να πούμε ότι η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπησέρχεται στην οργάνωση αυτή των εθνικών κρατών μελών. Άκουσα λοιπόν τα σχόλιά σας κυρία Περέ και είπατε ότι η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση είναι κάτι το αρνητικό σε κάποιες περιπτώσεις ε, κινούμαστε προς πολιτική κατεύθυνση με τη χρήση των όρων αυτών και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να το κάνουμε στο θέμα του νερού. Το θέμα λοιπόν ποιο είναι. Κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχει μία πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας νερό και μάλιστα σε λογικές τιμές. Το πώς αυτό θα το διοργανώσουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επαφίεται, θεωρώ, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Εγώ προσωπικά το λέω ανοιχτά. Είμαι από μια χώρα όπου είναι στα δημόσια χέρια η υδροδότηση. Και μιλάμε για το ποσοστό 90%. Άρα εγώ υποστηρίζω αυτό το δημόσιο μοντέλο, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και θα πρέπει εδώ να μείνουμε στα όρια που μας επιτάσσουν οι συνθήκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ, λέει ο κύριος Γκρούτ, που τηρήσατε και το όριο. Ναι, από πλευρά, ο κύριος Λάινεν, ο, από πλευρά των σοσιαλδημοκρατών, να ευχαριστήσω ιδιαίτερω τους οργανωτές της Ευρωπαϊκής αυτής πρωτοβουλίας των πολιτών. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα του νερού. Όλοι χαρήκαμε που τόσο, ένα τόσο ε, σημαντικό θέμα ήταν στο επίκεντρο αυτή του εργαλείου και γνώρισε τόσο μεγάλη ε, επιτυχία με την ε, αντίδραση του Μισελ Μπαρνιέ σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη στις σχετικές οδηγίες και με την ακρόαση εδώ πέρα που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σαφές ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία θα είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα καλέσουμε και στο μέλλον. Είμαι λοιπόν ε, Συχνά λοιπόν ψάχνουμε να δούμε που κινούνται τα ευρωπαϊκά κινήματα και χαίρομαι λοιπόν που με, ευρωπαϊκό αυτό, με την Ευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία για το νερό βλέπουμε ε, μια κίνηση, ένα κίνημα ευρωπαϊκό από κάτω προς τα πάνω και χαίρομαι γιατί θεωρώ ότι έτσι μπορεί να καταλαγιάσει αυτή η σκεπτικότητα από πλευρά του κόσμου γιατί ο κόσμος θα έχει την εντύπωση ότι μπορεί να συμμετάσχει πραγματικά σε κάτι. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλές νομοθεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα όμως ότι αφορά την εφαρμογή. Εγώ μένω κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, με το Λουξεμβούργο και ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά τέτοιες διαμεθοριακές περιοχές ε, είναι όλο και πιο σημαντικό να διευκρινίζουμε. Το 2027 Το 2015 έχουμε θέσει ως έτος στόχο σε ό,τι αφορά αυτά τα ρηχτά ζητήματα. Έχουμε ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι αφορά την κατασπατάληση του νερού. Πολύ νερό λοιπόν σπαταλάτε στη γεωργία, στα νοικοκυριά, στη βιομηχανία. Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ παραπάνω πράγματα και με τα περιφερειακά μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι το νερό θα πρέπει να περάσει και να βρει το τη θέση του και σε όλε τι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Γιατί ξέρετε δεν είναι ένα σύνηθε αγαθό, είναι το υπαριθμόν ένα αγαθό. Και αυτό θα πρέπει να είναι σε δημόσια χέρια και όχι να χρησιμοποιείται ιδιωτικά για κερδοσκοπία. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Γιολάινεν, ο κύριο Κρι Ντέιβι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι η ποιότητα της δημόσιας υδροδότηση πόσιμου νερού πρέπει να είναι πάντοτε υψηλή ποιότητα. Νομίζω και τα αποχαιρετικά συστήματα χρειάζονται νέε επενδύσει σε πολλέ περιπτώσεις, αλλά Σίγουρα πρέπει να έχουμε τα καλύτερα δίκτυα στην Ευρώπη. Πάντω, ιδιωτικοποιήθηκε πριν από 25 χρόνια σε εμά το σύστημα υδροδότησης και ε, αποχέτευση. Μάλιστα, με του ε, φιλελεύθερου ε, να γιγούνται αυτή τη μεταρρύθμιση, αντιταχθήκαμε τότε, όμω βρισκόταν στην καρδιά της ε, μεταρρύθμισης στο δημοσίου τομέα και των κοινοφελών υπηρεσιών. Ένα νέο σύστημα λοιπόν δημιουργήθηκε και τώρα έχουμε πολλέ νέες ιδιωτικέ εταιρείε ενώ μόνο ένας κρατικός ρυθμιστής που πρέπει να προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, ελέγχει τις εταιρείες αυτές, τις οποίες πρέπει να πιέζει να κάνουν επενδύσεις, να περιορίζουν τα κέρδη τους εάν δεν γίνονται επενδύσεις και να επιβάλλει πρότυπα ποιότητας καθώς και να προστατεύει αυτούς από τους οποίους μπορεί να κοπεί η υδροδότηση οποιαδήποτε άλλη πρόσβηση. Είναι ακριβό πάντως το σύστημα της υδροδότησης. Είναι δαπανηρό το σύστημα της αποχέτευσης, το να παράσχουμε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό. Είναι αλήθεια αυτό και οι χρήστες του νερού πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Και πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η παροχή του νερού είναι τόσο ε, αποτελεσματική και επαρκής όσο το δυνατό περισσότερο μάλιστα. Η εμπειρία μου στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι γίνεται αυτό να το παράσχει και ο ιδιωτικός τομέας, αρκεί να υπάρχει και ένας ρυθμιστής από την πλευρά του κράτους, δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος, και να βεβαιώνεται ότι τα συμφέροντα αυτά καλύπτονται και φροντίζονται επαρκώς. Ο από τους Πράσινους. Ευχαριστώ και φυσικά θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μπερέτ Περέτ ε, για την πρωτοβουλία και για την τεράστια επιτυχία που είχε, κάτι που δείχνει την τεράστια σημασία αυτού του θέματος, ιδιαίτερα για τους ε, πρασίνους. Και με αυτή την άποψη μπορούμε να ε, υμνήσουμε όλοι και να γιορτάσουμε αυτή τη στιγμή της συμμετοχικής δημοκρατίας. Το θέμα όμως είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και την επιτυχία της, αλλά από εδώ και πέρα τι μέλη ενέστε. Μέχρι στιγμής ήταν κάπως απογοητευτικός ο κύριος Εύτσοβιτς. Δεν θέλω να σας χαλάσω το κέφι, αλλά υπάρχουν ε, κάποια σημαντικά θέματα. Είπαμε ότι είναι γιορτή της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ωραία αυτά, αλλά στην πράξη τι σημαίνουν όλα αυτά. Και όπως ο συνάδελφος ε, συμφωνώ ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά σε τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη αποφασίζουν. Ή το ένα όμως ή το άλλο. Αν συμφωνήσουμε ότι πρόκειται για ανθρώπινο δικαίωμα, τότε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, τι προτείνε για το, κλιμα... για το κλιματικό αναλογό για το 2030, για το σχιστολιθικό αέριο, τίποτα. Αν έχουμε μια πηγή ενέργειας που θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού είναι το σχιστολιθικό αέριο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία δράση. Γιατί, αν θεωρείτε το νερό σημαντικό θέμα και το θεωρείτε ανθρώπινο δικαίωμα και αν θέλετε να, όλοι να έχουν πρόσβαση σε πόσιμο καθαρό νερό σε λογικές τιμές, θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Και τι γίνεται με την ιδιωτικοποίηση. Επίσημα ε, μας είπε ο κύριο Σεφτσοβιτς ότι δεν εμπίπτει σε αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν δείτε όμως ε, στα, Τρόικε και το μνημόνιο συνεννόησης ε, Τρόικας και, και δεν αναφέρεται τίποτα. Όμως στην έκθεση προόδου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι μέλος της Τρόικα ζητά την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση το τομέα του τομέα σύντατος της Πορτογαλίας. Άρα ε, παροτρύνει σε ιδιωτικοποίηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πορτογαλία για παράδειγμα. Άρα δεν είναι και αυτό που είπατε ότι δεν πιέζεται για ιδιωτικοποίηση. Πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο, αντί να μιλάμε όλοι για ύμνους, επένους, εγκόμια και γιορτές, καλύτερα να περάσουμε σε πρακτικά θέματα πολιτικής. Ευχαριστώ. Next <coughs> E η κυρία Σόζα εκ μέρου τη ΚΟΕ. Ευχαριστώ ε, όλους. Ε, καλησπέρα σα, εκ μέρου τη ΚΟΕ. Ήθελα να ευχαριστήσω όλου του διοργανωτέ αυτή τη πρωτοβουλία, όσου αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα εδώ, όλε και όλου που επέτρεψαν να γίνει αυτό σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό και η ομάδα μου προφανώ συμφωνεί με τι διεκδικήσει τη πρωτοβουλία των πολιτών Δηλαδή χρειάζεται υδροδότηση και αποχέτευση που να αγνωριστεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πρέπει να προστατεύεται δεν μπορεί να θεωρείται ένα εμπορικό αγαθό. Δεν είναι ένα εμπόρευμα σαν τα άλλα ε, αυτή η υπηρεσία. Και δεν μπορεί να είναι ιδιωτικό, ε, ιδιωτική διαχείριση του, παραμείνει στο χώρο του δημοσίου δικαίου. Πρέπει το κράτος να εξασφαλίζει το δικαίωμα και την πρόσβαση στο νερό και την αποχέτευση σε όλους και όλες. Όπω είπε ο συνάδελφο Ζίμπερ, δεν μπορούμε να παραμβούμε στι αποφάσει και τι επιλογέ των κρατών μελών. Να θυμίσω όμω και το είπε μόλις ο συνάδελφος ε, από τους Πρασίνους ότι η Τρόικα ε, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιβάλλουν τέτοια προγράμματα λιτότητα στα κάτι μελη που οι πολίτε δεν ε, έχουν πρόσβαση στο νερό σε πολλέ περιπτώσει. Στην χώρα μου, την Πορτογαλία, συμβαίνει αυτό. Και το ίδιο και στην Ελλάδα, όπου η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την υδροδότηση στην Αθήνα. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ δείχνει ότι σε 22.000 κατοικίες έχει κοπεί η υδροδότηση επειδή τα άτομα αυτά δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και μόνο 6.000 αποκαταστάθηκαν από αυτές που είχαν κοπεί. Ε, τις παροχές νερού. Θα πρέπει λοιπόν η Τρόικα να ξανασκεφτεί τη λιτότητα που επιβάλλει στους Ευρωπαίους πολίτες. Ιδάλλως το δικαίωμα στο νερό θα είναι μια πολύ ωραία ρητορική επινόηση αλλά δεν θα έχει καμία υλοποίηση στην καθημερινότητα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και έτσι ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο των ε, ερωτήσεων και των δηλώσεων για το θέμα αυτό και λοιπόν τώρα έχουμε την Επιτροπή των Πολιτών. Έχετε 10 λεπτά για να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακούσαμε. Κυρία Περέτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν δεν έχετε αντίρρηση θα ήθελα να δώσω το λόγο και στα μέλη της Επιτροπής των Πολιτών, ώστε να μην μονοπολίσω εγώ το λόγο. Θα ήθελα πάντως, για να ξεκινήσουμε αυτό το διάλογο, να πω ότι είναι σαφές ότι αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα στο νερό δεν θα πρέπει να μείνει ευσεβής πόθος θα πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί, να δοθεί σε αυτό το δικαίωμα σάρκα και οστά. Σήμερα το πρωί υπενθύμησα στον Επίτροπο Σεύτσοβιτς ότι αυτό που ουσιαστικά ζητούμε και διεκδικούμε και μπορεί να είμαστε ουτοπιστές και θεροβάμονες, αλλά αυτό που ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να αναθεωρήσει την ομοθεσία της. Γιατί έγιναν κάποια πράγματα σε επίπεδο της οδηγίας για το νερό, σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση, μπορεί να μην μας ικανοποιούν πλήρως, γιατί κατά τη γνώμη μας ύψιστη προτεραιότητα είναι το νερό ως θεμελιώδες δικαίωμα και αυτό θα πρέπει να φανεί, να κατοχυρωθεί και να διατρανωθεί σε μια γενική οριζόντια νομοθεσία που θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες οδηγίες. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ανελίνα Αρστρομ από τη Σουηδία, που επίσης είναι μέλος της Επιτροπής των Πολιτών. Ανέλη, παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Πολύ συχνά έχει κάνει την εντύπωση ότι μόνο στα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με το νερό. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι η πρόσβαση στο πόσιμο είδωρ είναι υπό απειλή. Ακόμη και σε χώρες που θεωρούσαμε ευημερούσες και σε πολύ καλή θέση. Να σας δώσω το παράδειγμα της χώρας μου, της Σουηδίας, όπου σε, πολλές, όπου σε πολλά σημεία του δικτύου το δίκτυο δεν λειτουργεί. Οι πλημμύρε είναι κάτι που θα πρέπει να μάθουμε να χειριζόμαστε στο μέλλον ω αποτέλεσμα των ε, κλιματικών αλλαγών. Εάν καταρρεύσουν τα δίκτυα υδροδότησή μα, αυτό θα είναι αποτέλεσμα τη κατάστασης που έχει δημιουργηθεί σήμερα. Επειδή σου ειδικέ εταιρείε νερού λόγου χάρη δεν έκαναν αρκετές επενδύσει εκεί που έπρεπε για να δημιουργήσουν νέα δίκτυα, για να ανανεώσουν ή να επισκευάσουν αυτά που υπήρχαν. Αυτή λοιπόν η απειλή είναι σημαντικότερη και πιο σοβαρή από αυτό που παρουσιάζουν ενδεχομένω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εάν θέλουμε ένα αηφόρο, ένα βιώσιμο σύστημα υδροδότησης και αποχέτευσης για το μέλλον, απαιτούνται οι κατάλληλες επενδύσεις και μάλιστα αμέσως στην Ευρώπη. Διαρκώς μιλούμε για την κρίση, για την ανεργία. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο κρίση και για να περιγράψουμε το τι συμβαίνει με τις κρατικές, με τις δημόσιες επενδύσεις στον τομέα του νερού. Χρειάζονται επενδύσεις τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Γιάν Βίλεν. Yes, thank you. Ε, ε, ναι, γεια σας. Είμαι μέλος και εγώ της Επιτροπής Πολιτών. Ε, θα ήθελα και εγώ να θίξω τα θέματα που έθεσαν δύο βουλευτές σε ό,τι αφορά την Τρόικα και την ιδιωτικοποίηση την οποία παρατηρούμε σε μια σειρά χωρών. Καταρχάς, η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών ε, ανησυχεί ιδιαίτερως για τις εξελίξεις αυτές. Η πρωτοβουλία μας δεν αναφέρει τίποτα για την ιδιωτικοποίηση, αλλά μας ανησυχεί το θέμα. Αυτό που μας λείπει είναι η αξιολόγηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς θα επηρεαστούν, πώς θα επηρεαστεί η πρόσβαση στο νερό που είναι ανθρώπινο δικαίωμα από την ιδιωτικοποίηση αυτό γιατί αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ως θεμελιώδες δικαίωμα, άρα δεν θα πρέπει να σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την ιδιωτικοποίηση των, της ιδροδότησης. Κάποιοι, αν δεν κάνω λάθος, ο βουλευτής από την ε, Αυστρία είπε ότι είναι θέμα κριτικής ευχαίρειας των κρατών μελών η ιδιωτικοποίηση. Αλλά οι εταιρείε υδροδότησης ε, στις χώρες ε, ε, αυστηρής ε, λιτότητας, είναι σαφές σε αυτές τις χώρες ότι υπάρχει και πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τρόικα να γίνει αυτό. Αν ε, δηλωθεί επίσημα ότι για παράδειγμα πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι συμφωνεί με την διαδικασία ιδιωτικοποίησης της επιδότησης στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, αυτό δεν ασκεί πίεση στις κυβερνήσεις. Άρα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να γνωρίζουμε ω το δικαίωμα την ιδρυοδότηση, αλλά αυτό δεν θα σήμαινε ότι θα έπρεπε αναγκαστικά να γίνουν μελετέ αντικτύπου για το πώ επηρεάζεται η πρόσβαση αυτή από την ιδιωτικοποίηση και πώ επηρεάζονται οι σχετικέ εξέλιξει. Είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν το ανθρώπινο δικαίωμα ιδρυοδότηση να εγκαθιδρυθεί στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αυτό να αλλάξει την οτροπία για τις εξέλιξεις αυτές. Ο βουλευτής από το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ιδιωτικοποίηση των εταιριών υδροδότησης. Και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε εκφράσει γνώμη για τις εξέλιξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ξανά και ξανά ο κόσμος μας λέει το εξή. Μας λέει ότι είναι αντιφατικές οι εκκλήσεις μας και τα αιτήματά μας. Λέμε λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να απελευθερωθεί, δεν θα πρέπει να διέπεται από τις ε, κανόνες της ενιαίας αγοράς ε, το θέμα της δεδότησης. Όχι, θέλουμε να μην απελευθερωθεί το θέμα αυτό. Ναι, αυτό ζητάμε. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου ακαθόδες αντιφατικό. Όχι, όχι. Όλες οι δημοσκοπήσεις ξανά και ξανά μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών καταδεικνύουν ότι ο κόσμος δεν θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός στις ε, ε υπηρεσίες Ακόμα και στον Ενωμένο Βασίλειο επί 20-25 χρόνια αυτό καταδεικνύουν οι δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν οτιδήποτε το αντιφατικό. Εκτός και αν έχει κανείς συμφέρον να προωθήσει την ιδιωτικοποίηση. Αλλά στους πολίτες, στο μυαλό του πολίτη, αυτό δεν είναι καθόλου αντιφατικό, καθόλου αμφιλεγόμενο. <laughs> Επόμενος υπάρχει κάποιος που να θέλει το λόγο από την Επιτροπή των, ε, της Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Μάλλον όχι, οπότε... Πρόεδρε, μπορούμε να προχωρήσουμε. Μάλιστα, έτσι ολοκληρώσαμε λοιπόν τον πρώτο γύρο και θα ήθελα να σα υπενθυμίσω σε ποιο κομμάτι βρισκόμαστε, σε ποιο τμήμα. Είμαστε στο θέμα της καθολικής πρόσβασης στο νερό και στις ε, υπηρεσίες αυτές για όλους. Το δεύτερο στη δεύτερη ενότητα. Έχουμε λοιπόν την κυρία, τη συνάδελφο κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και χαίρομαι για την διοργάνωση αυτής της συζήτησης με βάση την πρώτη αυτή πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών που αποτελεί μια καινοτομία της Ιθήκης Λισαβόνας. Πρωτοβουλία αφορά το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό αλλά μην ξεχνάμε ότι η πρόσβαση στο νερό είναι απαραίτητη και για την υλοποίηση άλλων δικαιωμάτων. Είναι απαραίτητο λοιπόν ε, και για την ε, ζωή, τη δημόσια υγεία, την ε, αξιοπρέπεια, την ευημερία. Είναι αναφυσβήτητα όλα αυτά. Έχω όμως κάποιες απορίες και προβληματισμό. Γιατί η συζήτηση αυτή με φοβίζει μήπως παρεκτραπούμε σε υπερβολικά ιδεολογικές συζητήσεις και ένα είδος αντιπαλότητας μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και αυτό αποσπάσει την προσοχή μας, αυτή η αντιπαλότητα, από την ανάγκη υλοποίησης πρόσβασης της πρόσβασης και προσπελασιμότητας του νερού για όλους, γιατί αυτό συμβάλλει και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εμπλακούμε στην απόφαση για τη διαχείριση. Είναι σημαντικό όμως και θεμελιώδες κάθε Ευρωπαίος πολίτης να έχει πρόσβαση σε ε, πόσιμο νερό και μάλιστα σε λογική τιμή, σε μια τιμή που μπορεί να πληρώσει, που θα είναι σε θέση να καταβάλει. Πάντως ε, πιστεύω ακράδαντα ότι η υλοποίηση του δικαιώματος αυτού στο νερό για όλους στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη μορφή του φορέα παροχής υδατός. Μπορεί να είναι και ιδιωτικός αυτός ο φορέας και δημόσιος. Το θέμα είναι οι κρατικές αρχές να έχουν τον έλεγχο και οι κρατικές αρχές να είναι πλήρως ελεύθερες να αποφασίσουν σε ποιο θα αναθέσουν την υπηρεσία της υδροδότησης, σε ένα δημόσιο ή σε ιδιωτικό φορέα. Ο έλεγχος πάντως παραμένει στις δημόσιες αρχές και θα πρέπει ακόμη και οι ιδιωτικοί φορείς να προσυπογράφουν τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και να αναγνωρίζουν το είδωρο ως ανθρώπινο δικαίωμα. Πάνω από 33% των ανθρωπίνων, των Ευρωπαίων πολιτών ε, έχουν πρόσβαση σε είδωρα ε, που το διαχειρίζεται μια ιδιωτική επιχείρηση. Ε, ακούσαμε όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει το Ινστιτούτο Thomas More ότι πολλά εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο είδωρα. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν, ποια είναι τα ακριβή στοιχεία και τα πιο αξιόπιστα. Γιατί φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά. Ευχαριστώ για τα δύο λεπτά. Ο Πίτερ Γιάρ, δύο λεπτά επίσης. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές. Ε, πραγματικά σήμερα μας βοηθάτε για μια πρώτη τέτοια ακρόαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φέρετε μια βάση για μια, ένα καλό πάτημα στην ευρωπαϊκή πολιτική και Όλοι ξέρουν, θα ξέρουν λοιπόν ότι αν θέλουν πραγματικά μπορούν να συμμετάσχουν. Αυτό λοιπόν καταδεικνύει πόσο σοβαρά παίρνουμε τα πράγματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω κι εγώ μια επιθυμία. Θα ήθελα η ακρόαση αυτή όχι μόνο να επιβεβαιώσει τις ήδη υφιστάμενες απόψεις και τοποθετήσεις. Όχι, θέλουμε να ακούσουμε, θέλουμε να θέσουμε ερωτήματα. Γι' αυτό λοιπόν να περάσω κατευθείαν στις ερωτήσεις. Να κάνω μια, μια μικρή παρατηρήση γιατί είμαι από μια περιοχή όπου προσπαθήσαμε και πιστέψαμε ότι όλα είναι στα δημόσια χέρια και τότε όλα θα πήγαιναν καλά και καμιά φορά βλέπουμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν ε, αντίθετα. Εγώ είμαι γενικά κατά της ιδιωτικοποίησης, αλλά να μην είμαστε αδιάλακτοι. Μία ερώτηση, το είπε σωστά ο συνάδελφος Ζέμπερ, ότι το η πρόσβαση για... στο νερό είναι ένα δικαίωμα για όλους και τώρα διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει να είναι και υψηλής ποιότητας και υγιεινό και σε λογικές τιμές. Με την απαγόρευση απελευθέρωση, τι καταλαβαίνετε εσείς, ε? απαγόρευση και ιδιωτικοποίηση, γιατί υπάρχουν διάφορα μοντέλα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν ας πούμε στη Γερμανία μοντέλα όπου οι δήμοι και οι κοινότητες εξακολουθούν να έχουν τη διαχείριση αλλά σε θέματα λειτουργικά ε, ανατίθεται στα ιδιωτικά χέρια και αυτό δεν είναι πάντα Και στη δική μου περιοχή έχουμε διάφορα μοντέλα ε, και σε ό,τι αφορά την δημοτική και την ιδιωτική διαχείριση και εγώ ως εξωτερικός παρατηρητής δεν βλέπω διαφορά ούτε στις τιμές ούτε στην ασφάλεια υδροδότησης. Αυτό απλά το διαπιστώνω. Φυσικά ε, αυτό που τονίζουμε ότι η απόφαση του Δήμου και των κοινοτήτων θα πρέπει να μείνει στα δημόσια χέρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο κύριος Μπαλτίνη είναι ο επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά από τους Σολδημοκράτε. Ευχαριστώ. Όλοι οι πολίτες χρειάζονται καθαρό πόσιμο νερό και καλό αποχετευτικό σύστημα. Το καθαρό πόσιμο νερό και το, η αποχέτευση είναι βασικά θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που θα πρέπει να εξασφαλιστούν με ζωστή ίδρυυση και αποχέτευση που θα πρέπει να είναι στοιχειώδεις δημόσιες υπηρεσίες. Και μάλιστα... Ε, ε, συνυπόγραψα μια διακήρυξη κατά της ε, ιδιωτικοποίησης των ε, τέτοιων δημόσιων αγαθών. Και μάλιστα κατάγομαι από μια χώρα που εγγυάται και εξασφαλίζει τους πολίτες τέτοιο πόσιμο νερό και δημόσιες υπηρεσίες ίδρυυσης, ενώ 80% των πολιτών υποφελείται από αυτό το σύστημα. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία «Το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα» γιατί θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να παροτρύνουμε τους νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαιτήσουν από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο και προστό σε τιμές είδωρ και αποχέτευση για όλους τους πολίτες και θα πρέπει να εκπίπτουν από του κανόνε τη δημόσια αγορά σε τομείς αυτής. Είναι σημαντική ε, και βασική αρχή και των σοσιαλιστών και δημοκρατών. Είναι απαραίτητο το δικαίωμα για τη ζωή. Κανένα ζωντανό πλάσμα δεν μπορεί να ζήσει στον πλανήτη χωρί ε, το απαραίτητο αυτό αγαθό. Ε, και επίση είναι σημαντικό για, τις, για το για το περιβάλλον. Τέσσερι όμω στου δέκα πολίτε στον κόσμο δεν έχουν τέτοια πρόσβαση ούτε καν σε τουαλέτε. Και δύο στου δέκα πολίτε δεν έχουν πρόσβαση στο νερό. Θα ήθελα λοιπόν να στείλουμε με βάση και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ε, την, την, την, ε, το μήνυμα αυτό και επίσης να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας για τους πολίτες μας που είναι πλημμυροπαθείς. Το ψήφισμα του 2010 των Ηνωμένων Εθνών 64-292 αναγνωρίζει ως ε, βασικό και θεμελιώδης δικαίωμα ανθρώπινο την πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση. Είναι σημαντικό λοιπόν η πρόσβαση στην ίδρυυση και την αποχέτευση για την υλοποίηση και των άλλων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνει το νερό ως δημόσιο αγαθό. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την, την πρόσβαση στις πηγές του νερού, γιατί για παράδειγμα και η Σλοβενία υποφελείται από τις δικές μας πηγές. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσει να υλοποιηθούν αυτά τα αναπαλωτήρια των ανθρώπινα δικαιώματα και να υλοποιηθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της ε, χιλιετίας. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης και της ε, διαίρεσης να γίνει το νερό στοιχείο σύνδεση μεταξύ των λαών και των χωρών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα έχω ε, την κυρία Σόσορ που ζήτησε το λόγο πάλι. Ευχαριστώ. Το θέμα που ανακύπτει είναι κατά πόσον το πόσιμο νερό στον 21ο αιώνα θα διαδραματίσει το, τον ίδιο ρόλο με το πετρέλαιο στον 20ο αιώνα. Και αν ε, αυτό όντω γίνει, το νερό θα έχει μεγάλη επιρροή σε αυτόν τον ε, αιώνα. Καλωσορίζω λοιπόν τη σημερινή πρωτοβουλία, καλωσορίζω και τι δηλώσει που έγιναν, γιατί με τον τρόπο αυτό ασκείται η άμεση δημοκρατία. Εγώ Είμαι από την Κροατία. Στην, ε, ε, είμαστε λοιπόν σε τέτοια θέση με την Νορβηγία και την Ισλανδία. Στην Κροατία το νερό ε, είναι δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο προστατεύεται ιδιαίτερο. Σε εθνικό επίπεδο ε, σκοπός μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση των αποθεμάτων. Αυτά δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν. Οποιαδήποτε απόπειρα ιδιωτικοποίηση θα αποτύχει παταγωδό στην Κροατία, αλλά ασφαλώ να έχουμε υπόψη και την επικουρικότητα. Γι' αυτό λοιπόν ρωτώ το εξή. Όντω, σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν επιλογή. Αυτή την εβδομάδα ζήτησα από την Επιτροπή να δραστηριοποιηθεί, να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης κατά των ε, ε, δύσκολων ε, ε, καιρικών συνθήκων στην Κροατία. Αυτή λοιπόν είναι η ερώτησή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών έχει αποδείξει ότι στον τομέα της υδροδότησης στην Ευρώπη Υπάρχει μάλλον μια κατάσταση που θα μπορούσαμε να την περιγράψουμε ως άναρχη. Σε ορισμένες χώρες ε, το κράτος αναλαμβάνει την ίδρυυση, ε, σε άλλες έχει ιδιωτικοποιηθεί η υπηρεσία αυτή. Στη δική μου τη χώρα η ίδρυυση ήταν στα χέρια του κράτους. Όμως, λόγω της προσχώρησής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγο πολύ εξαναγκαστήκαμε να ξεκινήσουμε διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση, διαδικασία ιδιωτικοποίησης μάλλον, της, του τομέα ίδρυυσης και συμμετείχαν και Γάλλοι, γαλλικές εταιρείες. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει σε δεκαπλασιασμό των προηγούμενων τιμών. Αυτό ήταν ιδιαίτερα επιβλαβές, ιδίως για όσους ε, είχαν ε, πρόσβαση στο αποχαιρετικό σύστημα και τώρα πια αποκλείονται από αυτό διότι δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία. Δεν μπορεί οι ιδιωτικοί επενδυτές ή εταιρείε να αφήνονται ελεύθερες, να κυνηγάνε το κέρδος που επιδιώκουν. Η πρόσβαση στο νερό είναι ένα θεμελιώδης δικαίωμα, ασχέτως του πώς εξελίσσεται και διαμορφώνεται η αγορά. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ντουιρό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας. Εγώ είχα μια ερώτηση που αφορά όχι τόσο πολύ την ε, παροχή νερού, την ίδρυυση ή το αν τα αποχητευτικά συστήματα θα ανατίθενται σε δημόσιες κρατικές αρχές ή σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά περισσότερο για το θέμα του καθαρισμού. Διότι για το θέμα του καθαρισμού ξέρουμε ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο, μεγάλο ιδίως στις μεγάλες ε, το να ασχολείται κανείς με το με τον καθαρισμό των υδάτων μιας μεγάλης πόλης είναι κάτι που έχει τεράστιο κόστος και όταν αυτό ε, ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες από τις δημόσιες αρχές ε, είναι πολύ δύσκολο να επιβάλλουν προτεραιότητες στους ε, ιδιωτικούς φορείς και είναι πολύ δύσκολο να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσει και επειδή το κόστος τελικά αναγκάζεται να το καλύψει ο καταναλωτής, να το πληρώσει με το λογαριασμό του. Έτσι λοιπόν γίνεται μια ιδιωτικοποίηση κάπως συγκεκαλυμμένη σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για συμβάσεις παραχωρητικές και με τις δημόσιες αρχές να αναθέτουν στις ιδιωτικές εταιρείες κάποια κάποιε αρμοδιότητε, κάποια καθήκοντα, τα οποία όμω δεν μπορούν να επιβάλλουν να τα φέρουν ει πέρα ιδιωτικέ εταιρείε, ακριβώ γιατί υποβαθμίστε το κύρο του. Ε, αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει από την νομοθετική πλευρά και τη ρυθμιστική. Να δούμε τις παγίδες των μορφών ιδιωτικοποίησης και της πρόσβασης σε ποιοτικό πόσιμο νερό για όλους και ιδίως για αυτούς που έχουν επισφαλή εισοδήματα παντού σε όλη την Ευρώπη. Πραγματικά ο καθαρισμός του νερού ε, και στα ε, στις περιοχές της Υπέθρου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά εκεί είδαμε ότι ε, οι εταιρείε που αναλαμβάνουν πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο κόστος να καλύψουν το οποίο τελικά με τους λογαριασμούς τους πληρώνουν οι καταναλωτές. Και αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Σας ευχαριστώ και έτσι ολοκληρωμήσαμε τη διαδικασία Catch the Eye και τώρα λοιπόν η Επιτροπή των Πολιτών θα πάρει το λόγο. Η κυρία Πέρε θα δώσει το λόγο στους ε, αντίστοιχου ομιλητέ ή στον περιγνώμονες. Ευχαριστώ κύριε Γκρότε. Θα ξεκινήσουμε την τελευταία ερώτηση. Γιατί έχουμε έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα αποχέτευσης. Που μπορεί όμως να απαντήσει και στη δική σας ερώτηση κυρία Τζουιρόν. Και μετά θα δώσω το λόγο στον Έρχαρτ και στον Γιάνν Βίλεμ και εγώ θα μιλήσω στο τέλος για τα θέματα δημοσίου ιδιωτικού φορέα. Ο Didier, από τη ΣΕΖΕΤΕ. Όντως, ε, ε, εργάζομαι σε μια εταιρεία αποχέτευσης. Δεν σημαίνει ότι είμαι εμπειρογνώμονος, αλλά έχω κάποια εμπειρία στο θέμα αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι είχαμε καθυστερήσεις δεκαετιών ολόκληρων για θέματα αποχέτευσης και τώρα καλούμαστε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα και αυτή την καθυστέρηση γιατί οι υποδομές είναι πολύ δαπανηρές και έχουμε την ευκαιρία και την ευκολία αυτών των ιδιωτικών επιχειρήσεων που ουσιαστικά μας προτείνουν έτοιμα αργοστάσια και για τις χώρες της περιοχής που έχουν καθυστέρηση είναι πιο εύκολο να περάσουν από αυτές τις ιδιωτικές ε, εταιρείες από το να αναπτύξουν το δικό τους ε, σύστημα δημοσίων υπηρεσιών. Θα μιλήσουμε ίσω και αργότερα για αυτό το θέμα τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων. Υπάρχουν όμω κάποιε δημόσιε κοινοφιλεί υπηρεσίε στη Γαλλία και φαντάζομαι και αλλού που έχουν τέτοια εμπειρία σε θέματα αποχέτευση ή καθαρισμού των λιμάτων και που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Γιατί οι κοινοπραξίε μεταξύ δημοσίων φορέων στην Ευρώπη δεν γίνονται τόσο εύκολα. Γίνονται περισσότερο με χώρες, σε χώρες του τρίτου κόσμου, στην Ινδία, στην Αφρική. Ενώ στην Ευρώπη φαίνεται ότι έχουμε δυσκολία με τέτοιου είδου συνεργασίε μεταξύ δημοσίων φορέων που θα μας επιτρέψει να απεξαρτηθούμε κάπως από τους ε, ιδιωτικούς ε, τελεστές, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και θα μπορέσουμε έτσι με συνεργασία μεταξύ δημοσίων τομέων να συμβάλλουμε σε, στη βελτίωση της, των υποδομών. Επίσης ε, θα πρέπει να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες είτε στο θέμα της υδροδότησης ε, ή στο θέμα της υποχέτευσης, να κρατήσουμε αυτό το κοινοφελή χαρακτήρα. Γιατί στη Γαλλία, από την Γαλλική Επανάσταση, ε, οι κοινότητε ήταν υπεύθυνε για θέματα υδροδότηση και αποχέτευση, Επειδή όμως ε, ιδιωτικοποιήσαμε του τομεί και τις υπηρεσίες αυτές ή έγιναν παραχωρήσει οι κοινότητε χάνουν όλο και περισσότερο αρμοδιότητες. Χρειαζόμαστε έναν γιατρό κατεπηγόντος, παρακαλώ. Is he a doctor or somebody else who can... Okay. Πώς υπάρχει κανένας γιατρός στην αίθουσα.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 So, Μάλιστα. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Der Betroffenen geht's jetzt Φαίνεται ότι το άτομο που είχε προβλήμα ε, πάει κάπως καλύτερα και τώρα μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε την ακρόαση. Η Επιτροπή των Πολιτών έχει πάλι λοιπόν το λόγο. Μπορείτε να συνεχίσετε από εκεί που διακόψετε πριν από λίγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Διντία Ντιμόν είχε ολοκληρώσει. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον Έρχαρτ. Ναι και ζήτησε το λόγο προηγουμένω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ε, Γερμανός εκπρόσωπος της ε, Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας αυτής και ζήτησα τη λόγο μετά την εισήγηση του κυρίου Γιάρ ο οποίος και μίλησε για την κατάσταση στην Ανατολική Γερμανία και σύγκρινε την κατάσταση με αυτά που επικρατούν στις Ευρωπαϊκού Δήμου και κοινότητε σήμερα στη Γερμανία. Θεωρώ ότι αυτές οι δομέ αυτή η σύγκριση δεν στέκει. Άλλε είναι οι δομέ, άλλε είναι οι συσχετισμοί. Οι δήμοι και οι κοινότητε αποφασίζουν το πώ θα οργανώσουν την αποχέτευση και την υδροδότηση. Όντως λοιπόν ένα τμήμα των ε, Δήμων στην Ανατολική Γερμανία έχουν και ιδιωτική ιδιοκτησία και διαπιστώσαμε ότι στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις αυτές, ε, σε, ό,τι αφορά τους μετόχους δηλαδή αυτούς, ε, τα, και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις τα τέλη υδροδότησης είναι χαμηλά. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τους γενικότερους όρους στις επιχειρήσεις αυτές, ε, η υδροδότηση κατά κανόνα διέπεται από τιμές οι οποίες είναι αρκετά πιο χαμηλές από ότι ε, στις περιπτώσεις της δημόσιας υδροδότησης 10 έως 15%. Άρα οι τιμές λοιπόν μπορούν να διατηρηθούν χαμηλές και παράλληλα να χρηματοδοτηθεί και με την ε, τα επιτόκια επί του κεφαλαίου, η ιδιωτική συμμετοχή. Αυτό να το έχουμε υπόψη σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς μετόχους. Τα πράγματα αυτά ήταν ακριβώς λοιπόν τα ίδια όπως και με τις αμυγός δημόσιες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ, Έρχαρτ. Ο Βίλεμ. Και μετά θα ακούσουμε τον Πέτρο και τον Τομάζο και τελειώνουμε από πλευράς μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως ένα προσωρινό συμπέρασμα, Πρόεδρε, για την ως τώρα συζήτηση, αυτό το γύρο, ε, σημειώνω ότι υπάρχει μια συμφωνία από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, διακομματική, όλοι οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων που ε, πήραν το λόγο εδώ μίλησαν και ανέφεραν τη στήριξή τους για το δικαίωμα όλων στο νερό και τα, τις υπηρεσίες και αποχέτευσης. Εάν σκεφτούμε λοιπόν ποιε είναι οι αντιδράσει των Ευρωβουλευτών προ τι διεκδικήσει των Ευρωπαίων πολιτών και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι εισακούονται ε, οι δικέ μα οι απαιτήσει και ότι τι αναγνωρίζουν. Είναι δια... πολιτική και διακομματική η υποστήριξη και συνένεση αυτή. Τώρα για τα θέματα της απελευθέρωσης, της ιδιωτικοποίησης, ο κύριος Γιάρ νομίζω έθεσε ένα πολύ άμεσο ερώτημα. Και αν διαβάσει κανείς πιστεύω τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις των ε, πολιτών, της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί, να μην απελευθερώσει τι υπηρεσίε ίδρυυση και αποχέτευση ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό θα θέλαμε να είναι κάτι που θα καταγραφεί και σε νομοθετική βάση. Ε, να μην είναι μια ανακοίνωση, ένα δημοσίευμα ή να θαυτεί κάπου σε κάποιο χρονοτούλαπο, αλλά να αναφερθεί ρητός στην κοινοτική νομοθεσία ότι η Ευρωπαϊκή αλλα να αναφερθει ρητο στην κοινοτικη δεσμεύεται να μην απελευθερώσει την υπηρεσίε ίδρυυση και αποχέτευση. Και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ω μέρο των εμπορικών τη συμφωνιών. Θα το ακούσουμε αυτό και στον επόμενο γύρο στη συζήτησή μα. Κάποιε φορέ υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ απελευθέρωση, ιδιωτικοποίηση. Η δική μα πρωτοβουλία ζητά πραγματικά σαφή δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αναλάβει πρωτοβουλίε για την απελευθέρωση των υπηρεσιών υδροδότηση. Μα ανησυχεί η ιδιωτικοποίηση, όπω είπαν και πολλοί ευρωβουλευτέ εδώ, και είναι, απαραίτητο το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ισχύει να ισχύει ώστε να αποτιμώνται σωστά τέτοιε καταστάσει. Και πάλι το ΟΗΕ έχει ένα πολύ σαφέ πλαίσιο αναφορά για του τρόπου με τους οποίους θα μπορούσαμε να εφαρμόζουμε το δικαίωμα αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πέδρο και μετά το Μάζο. Ευχαριστώ. Ε, αναφέρθηκε πως είναι ιδεολογικό το πρόγραμμα. Δεν είναι, κακό, δεν είναι κακιά, κακή ιδεολογία, ούτε η ιδεολογική πολυμορφία, αρκεί να υπάρχει σεβασμός. Οπότε από αυτήν την άποψη είμαι ήσυχο. Δεν είναι όμως μόνο θέμα ιδεολογικό. Όταν πριν από τρεις μέρες είπαμε στην Ισπανία ότι 200 ε, ε, οικογένειες ε, στο Χερές de la Frontera, εκεί που γίνεται το τσέρι το Χερές, είδαν να κόβεται το νερό τους. Και έχουμε πια κάνει κάποιους λογαριασμούς και λέμε, βλέπουμε ότι σε χιλιάδες οικογένειες έχει κοπεί το νερό. Ε, και μου λέτε, it's up to you, από εσάς εξαρτάται. Το επιτρέπει η Ισπανική κυβέρνηση. Δίκαιο είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στην Ισπανική κυβέρνηση ή στην Πορτογαλική κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι θέμα ιδεολογία αυτό, είναι κάτι παραπάνω. Όταν έγινε διαβούλευση με τους Ιταλούς, ήταν 30 εκατομμύρια Ιταλοί. Φαντάζομαι να ήταν πολύ και δεξιοί και αριστεροί. Δεν ήταν θέμα ιδεολογίας, είναι, θέμα ανθρωπιστικών αρχών. Είμαι καθηγητής οικονομίας, μπορώ να σας δώσω οικονομικά στοιχεία. Έχουμε από την πατρίδα μου 20 χρόνια ε, εμπειρία ιδιωτικοποίησης. Στην Αλμοθάρα 100.000 ε, το επίσημο κόστος ε, για όλα, για την απόσβεση του κεφαλαίου διαχείρισης 0,15 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, καρτούχα. 25 χρόνια ιδιωτική εταιρεία. 0,41 το κόστος για το κυβικό μέτρο, τριπλάσια τιμή δηλαδή. Επίσης έχουμε σχέδιο αποχέτευσης στην αραγών, 1,3 ε, το κυβικό μέτρο, σχεδόν δεκαπλάσιο το ποσό. Και τελευταία ιδέα, αφήνουμε ελευθερία και διακριτική ευχαίρεια στα κράτη-μέλη. Εντάξει, να αφήσουμε ελευθερία στις ε, αρχές. Ερωτώ λοιπόν, μπορούμε να αφήσουμε ε, και την ελευθερία και στους πολίτες, να διαλέγουν και οι πολίτες, γιατί εκεί που έγινε διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες, σε δημοψήφισμα ήταν μαζική συντριπτική πλειοψηφία. Φοβόμαστε να κάνουμε διαβούλευση με τους Ευρωπαίους πολίτες μήπως. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκαν ε, ε, οι απαντήσεις των ερωτήσεων από πλευράς της Επιτροπής Πρωτοβουλίων και τώρα λοιπόν το λόγο έχει η Κυρία Μπένιγκ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλου. Ήθελα και εγώ να πάρω μέρο στη συζήτηση και να συμφωνήσω με του ομιλητέ που είπαν ότι είναι πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ σήμερα ω μέρο αυτή τη πρώτη Ευρωπαϊκή ε, Πρωτοβουλία των Πολιτών και με τι απαιτήσει αυτέ για το δικαίωμα στο νερό. Να θυμίσω ότι είμαστε εδώ, εγώ τουλάχιστον είμαι εδώ, για να δώσω κάποιε απαντήσει για τι περιβαλλοντικέ συνιστώσεις αυτής της πρωτοβουλία. Άκουσα πολλά για την εσωτερική αγορά και τη διάσταση αυτή, αλλά θα το αφήσω στους συναδέλφους που θα πάρουν μέρος στον επόμενο γύρο. Στη διεθνή συνιστόσα, τη συνιστόσα την εξωευρωπαϊκή. Να σας δώσω κάποιες απαντήσεις για την περιβαλλοντική πτυχή. Πιστεύουμε και συμφωνούμε ότι είναι ε, καθοριστικό το νερό για την ανθρώπινη ζωή και υγεία και είναι ένας φυσικός πόρος απαραίτητος και για την οικονομία μας. Γι' αυτό η διαφύλαξη και η προστασία των υδάτινων πόρων είναι βεβαίως ζωτική σημασία και ακρογωνίως λήθος της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική αυτή ε, ήδη έχει ληφθεί υπόψη από δεκαετίες με την οδηγία για το πόσιμο νερό, για τα αστικά λίματα ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και ασφαλείς υπηρεσίες αποχέτευσης. Επίσης υπάρχει η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, που προβλέπει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείριση των υδάτινων πόρων. Τώρα, για κάποιου αριθμού για όσου ζήτησαν αριθμητικά στοιχεία, να πω ότι βάσει των πρόσφατων δεδομένων που διαθέτουμε, κατά μέσο όρο 95% του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πρόσβαση στο νερό μέσω της, του δημοσίου δικτύου υδροδότησης και ο βαθμό συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερό που συζητούνται από τι οδηγίε είναι υψηλό πάνω από 90% κατά μέσο όρο. Για τα συστήματα καθαρισμού των νερών και τη διασύνδεση φτάνουμε το 85% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 94% για την διαχείριση των αστικών λιμάτων από τις περιοχές που καλύπτονται από την οδηγία για τα διαχείριση των αστικών λιμάτων. Σωστά συλλέγονται και το 80% του νερού που παράγεται ε, υπόκειται στη σωστή επεξεργασία βάσει τη οδηγία για τα αστικά λύματα. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε διαφορέ ω προ τον ε, βαθμό συμμόρφωση μεταξύ των κρατών μελών, γιατί υπάρχει και ένα έλλειμμα ε, υλοποίηση, μεταφορά στα νέα κράτη-μέλη. Βεβαίω λοιπόν πρέπει να βελτιωθεί η υλοποίηση καθώ και η συμμόρφωση με τα συστήματα συλλογή και επεξεργασία του νερού, όμω ήδη υπάρχει ένα βαθμό βελτίωση ε, επιτάχυνσης της πρόοδου στα νέα κατημέλη λόγω της σημαντικής οικονομικής στήριξης από τα διευθυντικά και ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, από το 2007 πάνω από 2,6 εκατομμύρια πολίτες ε, είχαν ε, καλύτερη παροχή ε, ποιοτικότερου νερού και 5,5 εκατομμύρια νερό διασυνδέθηκαν με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης των αστικών λιμάτων. Μεταξύ του 2007 και το 2013 η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε στα συστήματα αυτά 22 δις ευρώ για τη βελτιωμένη υδροίδρευση και αποχέτευση. Όσο και τα παλιά κρατημέλη και το βαθμό συμμόρφωσης, ιδίως για τις διατάξεις σχέση με την ε, επεξεργασία των αστικών λιμάτων. Υπήρχαν και κάποιες ε, διαδικασίες ε, επιβολής, αλλά και υποστήριξη το, της χρηματοδότησης. Όπως απέδειξε το blueprint, το αποτύπωμα του 2012 για το νερό. Η διαδικασία που ακολουθήσαμε ως τώρα, μέχρι τώρα, ως τώρα ήταν επιτυχής και γι' αυτό θα εξακολουθήσει και στο μέλλον. Βεβαίως χρειάζονται περαιτέρω βελτιώσεις. Υπάρχει τέτοιο περιθώριο, γι' αυτό ήδη έχουμε ε, προγραμματίσει κάποιες δράσεις από το ε, blueprint του 2012 και με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Πρέπει να δώσουμε προσοχή στην καλύτερη ποιότητα του πόσιμου νερού για τους μικρούς παροχής, ιδίως σε περιοχές της υπαίθρου και πιο απομονωμένες περιοχές. Επίσης, όπως υπόθηκε εδώ, θα πρέπει να ενισχύσουμε τις επενδύσεις για την ε, οικοδόμηση σχετικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ίδρευσης, κυρίως στα κράτη-μέλη της Ανατολικής Ευρώπης. Και πολύ σημαντικό, θα πρέπει να ε, συντηρήσουμε διαχειρίσουμε σωστά τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον. Επίσης θα πρέπει να τονώσουμε την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών μέσων όχι μόνο για να έχουμε καθαρό νερό αλλά και για να έχουμε νερό που θα είναι αξιοποιήσιμο και θα σέβεται την ανάγκη διαφύλαξης των φυσικών μας πόρων. Εδώ σωστά αναφέρθηκε το θέμα της απόσβεσης, της ανάκτησης του κόστους και στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα υπάρχει μια τέτοια διάταξη ότι η αρχή αυτή ε, ανάκτησης του κόστους θα πρέπει να είναι μια αρχή που να διέπει τα συστήματα διαχείρισης ε, του νερού, ίδρευσης δηλαδή, από τα κάτι μέλη. Ε, επίσης θέλουμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση των καταναλωτών και βαθμό με, την οποία, με τον οποίο παρέχονται όλες αυτές οι υπηρεσίες με διαφάνεια προς τους πολίτες. Έναντι όλων αυτών των προκλήσεων έχουμε ήδη προβλέψει κάποιες δράσεις, ε, ορισμένες σε εξέλιξη και όπως είπα το να βελτιώσουμε τη διαχείριση των δεδομένων μας και τα συστήματα ενημέρωσης για να ενισχύσουμε το κεφάλαιο γνώση που διαθέτουμε για όλε τι διαστάσει που σχετίζονται με το νερό είναι σημαντικό. Μαζί με τα κράτη-μέλη έχουμε προγράμματα υλοποίηση με συγκεκριμένα ορόσημα, επενδυτικά προγράμματα και προτεραιότητε με δυνατότητε χρηματοδότηση. Η ποιότητα του νερού για του μικρού παροχή είναι κάτι που το βλέπουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη διαθέτουν ήδη ένα πρόγραμμα, για τις δράσεις, ένα πρόγραμμα πλαίσιο για τι δράσει του, μαζί με συγκεκριμένε κατευθυντήριε γραμμέ, με βέλτιστες δράσει για να βελτιώσουν ακριβώς το σύστημα των μικρών παρόχων. Και η κοινοτική νομοθεσία εξετάζεται προς αναθεώρηση. Για παράδειγμα η οδηγία για τις ε, προτερε... ουσίες προτεραιότητες που πρόσφατα επικαιροποιήθηκε ή η οδηγία για τους υδροφόρους ορίζοντας που πρόκειται να επικαιροποιηθεί καθώς και η οδηγία για το πόσιμο είδωρ. Είναι κάτι που βρίσκεται στη διαδικασία της εξέτασης των διατάξεων παρακολούθησης και μεταφοράς. Τέλος, ε, να πω ότι προφανώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή και του κοινού, των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για το νερό ήδη προβλέπει μηχανισμό για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ούτως ή άλλως. Είμαστε πλήρως συμμορφούμενοι με την σύμβαση του όρχους και ε, οι, περιβαλλοντικές, μελέτες περιβαλλοντικού δικτύπου για όλα τα στάδια του προγραμματισμού είναι κάτι που ε, ήδη έχει μελετηθεί και εγκρίθηκε κιόλα από το Ευρωκοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να πω εν είδη συμπεράσματο ότι οι δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το νερό και την αποχέτευση ε, τα τελευταία χρόνια έχουν επιτρέψει την πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίε στη μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν ακόμη προκλήσει μπροστά μα για το μέλλον, αλλά τι αντιμετωπίζουμε σε συνεργασία και σε διαβουλεύσει με τα κάτι μελη και του ε, δημόσιου φορεί, ε, καθώ και του ενδιαφερομένου, προκειμένου να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την κοινωτική νομοθεσία για τα ύδατα και να υπάρχει πλήρη πρόσβαση όλων στο δίκτυο ίδρυυση και αποχέτευση. Ευχαριστούμε. Και τώρα λόγο στην κυρία Νόστρομ για συμπεράσματα από τον πρώτο μας γύρο. Eh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή και πολλέ και ενδιαφέρουσε οι απόψει που ακούστηκαν. Νομίζω ότι γενικώ όλοι συμφωνούμε ότι είναι τεράστια η πρόκληση προκειμένου να ανταποκριθούμε σε όλες τις πτυχές του θέματος. Είναι ενδιαφέρον ωστόσο το ότι διαπιστώνουμε ότι πολλά έχουν ήδη γίνει, αλλά φυσικά πολλά ακόμα έχουμε μπροστά μας, γιατί πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση η διαρκής πρόσβαση στο νερό. Δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνάμε συζητήσαμε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μου δόθηκε η εντύπωση ότι ασχολούμαστε πιο εντατικά με τα θέματα αυτά. Πρόκειται όμως για ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα στην πρόσβαση στο νερό και ως τέτοιο θα πρέπει να ε, καταξιωθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητέ για τις παρουσιάσεις τους για τον πρώτο γύρο και τώρα θα περάσουμε στον δεύτερο γύρο σε ό,τι αφορά την ε, ε, καθολική πρόσβαση στο νερό και στην υδρατότηση για όλους. Θα αλλάξουμε λοιπόν τα μέρη του πάνελ και θα έρθουν καινούργιοι ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε με ένα μέλος της Επιτροπής των Πολιτών, τον κύριο Πέδρο Αρόχο. Έχετε πέντε λεπτά κύριε Αρόχο για να μας κάνετε την παρουσίαση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζούμε ένα πολύ δραματικό παράδοξο στον κόσμο. Η παγκόσμια κρίση για το νερό λαμβάνει χώρα στον πλανήτη του νερού, στο γαλάζιο πλανήτη. Έχουμε μια κρίση που δεν είναι τόσο πρόβλημα ασπάνητος νερού, αλλά είναι η απόρρια τριών κεφαλαιοδών λαθών. Το πρώτο λάθος, η πρώτη κρίση, είναι η κρίση βιωσιμότητας που προκαλέσαμε στα θαλάσσια και στα συστήματα τα οικοσυστήματα μας των υδάτων. Επίσης, η κρίση της ανισότητας και της ένδυας εξαιτίας του κοινωνικο-οικονομικού συστήματός μας που είναι τελείως ανήθικο. Και τέλος, είχαμε την κρίση της, της διαχείρισης των υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης εξαιτίας των πιέσεων ιδιωτικοποίησης που μετατρέπουν τους πολίτες μας σε απλούς πελάτες, περιθωριοποιώντας τους πιο ευάλωτους και φτωχότερους. Οπότε η έλλειψη βιωσιμότητα, η φτώχεια και η έλλειψη δημοκρατία ουσιαστικά είναι οι ρίζε του κακού, οι ρίζε αυτή τη κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία πλαίσιο για το νερό, στο μέτρο που αντιμετωπίζει το πρώτο από τα λάθη και το πρώτο από τι κρίσει που ανέφερα, ασκεί μια πολύ σημαντική ηγετική θέση και διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ε, υδάτινων οικοσυστημάτων και των σημαντικών αξιών και λειτουργιών που διακυβεύονται. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε την κατάλληλη νομοθεσία που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές αξίες που σχετίζονται με τις χρήσεις ε, και τις υπηρεσίες του νερού και τις παραγωγικές και τις υπηρεσίες ε, ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ε, δεν αντιμετωπίσαμε τα βασικά προβλήματα της φτώχειας και της ανισότητας, ούτε τις αντιφάσεις που προέκυψαν από την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ουσιαστικά λοιπόν ξεριζώσαμε την ψυχή, την κοινωνική ψυχή της νομοθεσίας μας και αφήσαμε σε κάθε κράτος μέλος να γεφυρώνει αυτό το κενό και να καλύπτει αυτό το χάσμα όπως μπορεί. Η, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών με το Right to Water, το δικαίωμα στο νερό δηλαδή, με σχεδόν 2 εκατομμύρια υπογραφές, ε, απαιτεί να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση για τις ε, διακυβευόμενες κοινωνικές αξίες για να εξεταστούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πολιτών αλλά με ηθικό πρίσμα με την αναγνώριση της πρόσβασης ε, σε, σε πόσιμο είδωρ και σε βασικές υπηρεσίες αποχέτευσης ε, και να αναγνωριστούν όλα αυτά ως ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνώρισε και η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ώστε να διαφοροποιήσουμε το ανθρώπινο δικαίωμα των 30-40 λίτρων το άτομο τη μέρα για πόσιμο νερό από το εύλογο δικαίωμα να χρησιμοποιεί κανείς νερό για να κατασκευάσει ε, χαρτί, να γεμίσει μια πισίνα ή να ποτίσει ένα κήπο. Πρόκειται για μια ηθική, κοινωνική και σε τελική ανάλυση πολιτική συζήτηση που επιτρέπει στην Ευρώπη να ανακτήσει την έγκλη τη ε, σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών και να ξεπεράσει την απλή μερκαντιλιστική εμποροκρατική λογική. Μια συζήτηση που θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε την ηγετική μας θέση που σήμερα την χάσαμε και που την ασκούν άλλες χώρες για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι η περιπλοκότητα των διακυβευόμενων αξιών σε θέματα νερού ξεπερνούν τις δυνατότητες αγοράς και η σύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τα δικαιώματα των ανθρώπων θα πρέπει να εξασφαλίσετε και οικονομική ε, οικουμενική συγγνώμη, πρόσβαση έρχεται σε κατάφορη αντίφαση με την εμποροκρατική λογική. Στο μέτρο που απαιτεί νέα ε, μοντέλα δημόσια και συμμετοχική διαχείριση και όχι μόνο δημόσια διαχείριση. Προτείνουμε λοιπόν να ενισχυθούν τα κριτήρια, οι στόχοι και οι αρχέ τη οδηγία πλαίσιο για το νερό για την βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων μας του ύδατος. Επίσης, να αναγνωρίσουμε επίσημα και πανηγυρικά την πρόσβαση σε πόσιμο νερό και στοιχειώδεις υπηρεσίες αποχέτευσης ως στοιχειώδε και ε, βασικό ανθρώπινο δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσία. Να θεσπίσουμε μια συμπληρωματική νομοθεσία θα συμπληρώνει την οδηγία πλαίσιο και θα λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές αξίες ε, γύρω από τις διάφορες χρήσεις του νερού, εξασφαλίζοντας ε, την ε, υπεροχή της πρόσβασης στο πόσιμο νερό και στην εποχέτευση ως βασικό, ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι η πολυπλοκότητα και η φύση αυτών των αξιών, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων απαιτεί την ε, λήψη υπόψη του γενικού συμφέροντος της κοινωνίας και των επερχόμενων ε, γενεών στο επίκεντρο της προσοχής για να εξασφαλιστεί αυτή η πρόσβαση σε ίδρυυση και αποχέτευση. Επίσης, για να εξασφαλίσω αυτήν την οικουμενική πρόσβαση που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών, θα πρέπει να προβλέψουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο και, μια, και ένα νέο μοντέλο δημόσιας συμμετοχικής διαχείρισης, ξεπερνώντας την λογική της αγοράς, αλλά ξεπερνώντας και τις αδυναμίες παροχημένων μοντέλων δημόσιας διαχείρισης. Όπως και οι υπηρεσίες της δικαιοσύνης δεν είναι αντικείμενο αγοραπολισίας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αγοραπολισίας και ελπίζω να συμφωνούμε σε αυτό και οι βασικές υπηρεσίες ίδρυυση και αποχέτευσης δεν θα πρέπει να υπακούν στην απλή λογική του κέρδους πέμπτο και τελευταίο στοιχείο. Από την θέση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει την παγκόσμια της ευθύνη και να προωθήσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα διεθνού συνεργασία που θα στηρίζεται στην αρχή τη αλληλεγγύη και όχι τη ε, κερδοσκοπία και θα στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών και φορέων και δεν θα ε, προωθεί συγκεκαλυμμένες ε, μορφές ιδιωτικοποίηση με βάση τις στρατηγικές της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται αναγνω... παγκοσμίω ως το ευρωπαϊκό μοντέλο ιδιωτικοποίησης ουσιαστικά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα περνάμε λοιπόν στον πατογύριο ερωτοπαντήσεων και θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλοι να τηρήσετε το χρονικό όριο γιατί έχουμε καθυστερήσει και λίγο. Θα ήθελα λοιπόν να έχουμε και χρόνο και στον τρίτο γύρο ρετοπαντήσεων α, και για τις παρουσιάσεις ασφαλώς να έχουν το χρόνο τους. Μισελ Στρίφλερ, εισηγήτρια για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δικαίωμα για το Νερό από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που μπορώ σήμερα να εκπροσωπήσω την Επιτροπή Ανάπτυξη αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση στα πλαίσια τη της τελείω πρώτη ε, πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολίτων. Το δικαίωμα υδροδότηση και αποχέτευση ε, το ω οικουμενικό δικαίωμα στα περισσότερα κείμενα του ΟΗΕ. Το να ε, διασφαλίσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό που δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες είναι ο 7 στόχος των στόχων της χιλιετίας και η έκθεση του ΟΗΕ του 2013 για το πόσιμο νερό αναφέρει ότι σε σχέση με το στόχους της χιλιετίας το 2010 ο στόχος για την ίδρυψη έχει βελτιωθεί στο 2010 10, ενώ θα πρέπει να βελτιωθεί το δικαίωμα στην αποχύτευση. Ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία εκτιμά ωστόσο ότι 780 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο πόσιμο νερό και 2,5 δι δεν έχουν πρόσβαση στην ε, αποχέτευση. Στην ε, Αφρική Νοτίο τη Σαχάρα ειδικίω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί στι χώρε, στι αναπτυσσόμενε χώρε μεγάλα προγράμματα για την παροχή αυτών των υπηρεσιών αξίας πολλών δις ευρώ. Η ποιότητα του πόσιμου νερού είναι πολύ σημαντική για την ε, επισητιστική ασφάλεια. Οι ξηρασίες και πλημμύρες μπορούν να οδηγήσουν σε μετατομίσεις πληθυσμών και να οδηγήσουν σε εντάσεις και διεκδικήσεις ή σειράξεις ακριβώς για το θέμα του νερού. Επίσης μπορεί να προκαλέσει ε, πραγματική σύγκρουση η διεκδίκηση του νερού ε, η παροχή πόσιμου νερού μπορεί να προλάβει ακριβώς μία σύγκρουση. Χρειάζεται λοιπόν δράση η οποία να εξασφαλίζει ποιότητα ε, και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ένας αριθμός των πολιτικών μας να ε, εκπονηθούν και να μελετηθούν ακριβώ με αυτό το στόχο. Η εμπορική και η ενεργειακή μα πολιτική θα πρέπει να λάβουν υπόψη του προβληματισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι αναπτυσσόμενε χώρε καθώ και του το ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός των φυσικών υδάτινων πόρων που δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα εδάφη μόνο για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή ζωοτροφών ή εμπορευομένων αγαθών που να είναι εμπορεύσιμα. Πρέπει να καλύψουμε και τι ανάγκε των τοπικών πληθυσμών. Επίση πρέπει να περιορίσουμε δραστικά τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου διότι οι κλιματικέ αλλαγέ θα περιορίσουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε αυτό το ζωτικό αγαθό, το νερό. Θα πρέπει οι ευρωπαϊκέ εταιρείε να ε, κληθούν να σεβαστούν τι υψηλέ απαιτήσει ποιότητα στον τομέα του νερού και στι αναπτυσσόμενε χώρε και να δίνουν ε, λόγο για τι επιδόσει του τομέα αυτό. θα πρέπει να γίνει ανάληψη ευθύνη και να συμβάλλουμε εμεί οι ίδιοι στο δικαίωμα πρόσβαση στο νερό στι αναπτυσσόμενε χώρε, χωρί να αγοράζουμε ε, προϊόντα τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη την προστασία αυτού του δικαιώματο και θα πρέπει να ενημερωνόμαστε καλύτερα. Διότι πολλέ φορέ αυτό που λείπει είναι η διαφάνεια. Με τι εκτιμήσει των ε, 1.800 παιδιών κάτω των 5 ετών που πεθαίνουν καθημερινά λόγω οξίας διάρειας από λόγους που έχουν να κάνουν με το νερό, την ε, αποχέτευση και την υγιεινή, αυτό δείχνει πόσο το νερό συνδέεται με το δικαίωμα στη ζωή, το πλέον θεμελιώδης δικαίωμα. Η διάσκεψη του ΡΙΟ συν 20 το 2012 είδα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβεβαιώνει την δέσμευσή της προς το δικαίωμα αυτό και την προστασία ε, της πρόσβασης σε πόσιμο νερό και αποχέτευση για όλους, σε όλες τις χώρε. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργαστούμε προ αυτόν τον κοινό στόχο. Να ευχαριστήσω του διοργανωτέ αυτή τη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία που συμπεριλάβαν το θέμα του νερού σε όλη τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη και ελπίζω όλοι να κάνουν το απαραίτητο ώστε να γίνει το δικαίωμα αυτό μια πραγματικότητα ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Με τα τέσσερα λεπτά με έκανα το καλύτερο μπορούσα. ευχαριστώ. Φιώνα Χόλμ είναι η επόμενη ομιλήτρια και έχει 1,5 λεπτό στη διάθεσή της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να απαντήσω σε αυτό που είπε η κυρία Σέφερ για τα θέματα αποχέτευση και ουσία αφορά τους στόχους της χιλιετίας, ότι δεν έχουμε, δεν ακολουθούμε τους στόχους μας. Η UNICEF είπε το 2010 ότι οι πλέον φτωχοί δεν είχαν κερδίσει το οτιδήποτε σε ό,τι αφορά θέματα αποχέτευση και αυτοί που λοιπόν δεν έχουν οποιαδήποτε ανάπτυξη είναι τα άτομα ε, τα πολύ φτωχά και τα άτομα με αναπηρία. Το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν είχαν καμία άλλη εναλλακτική από το από το να φοντεύουν σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά ε, χαρακτηριστική ένδειξη και η διάρκεια λοιπόν θερίζει και οι σχετικές μολύνσεις ε, ε, επηρεάζουν 400 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό φυσικά έχει τον αντίστοιχο αντίκτυπο και στην εξέλιξή του υπάρχει και ο περιβαλλοντικός ε, αντίκτυπος γιατί οι εκαθαρσίες οι ανθρώπινες εισέρχονται στα, στα, στα υπόγεια δίαιτα, και το 90% των ε, αποχετεύσεων στις φτωχές χώρες καταλήγει σε ποτάμια και ποταμούς και λίμνες. Χρειαζόμαστε λοιπόν τέτοιες τεχνικές για την διαχείριση των αποβλήτων. Χρειαζόμαστε να διασφαλίσουμε ότι το πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015 το οποίο προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα λάβει υπόψη σοβαρά την αποχέτευση. Τι κάνετε λοιπόν ερωτώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παραγωνιστεί αυτός ο στόχος της αποχέτευσης ότι αφορά το πλαίσιο για τους στόχους μετά το 2015. Ευχαριστώ. Ο κ. Χρυσόγελος από τους Πράσινους έχει το λόγο. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, σίγουρα μιλάμε για τους στόχους της χιλιετίας και για την αναγνώριση του δικαιώματος ε, πρόσβαση στο νερό, στο καθαρό νερό και στην αποχέτευση σαν βασικό και οικουμενικό δικαίωμα. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν πώς αυτό στην πράξη θα εφαρμοστεί κυρίως μέσα από τις αναπτυξιακές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αλλά ε, και μέσα από τις συμφωνίες με τρίτες χώρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η κρίση ή προβλήματα οικονομικά να μην προωθούν τελικά ε, πολιτικές ιδιωτικοποίησεις. Είδαμε και στην Κροατία αλλά και στην Ελλάδα με αφορμή την κρίση την οικονομική να επιβάλλονται όροι για ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών νερού ε, θα θέλαμε να το διαψεύσει η Κομισιόν και επίσημα ότι αυτά που προωθούνται δεν είναι κάτι το οποία επιβάλλονται από την ίδια την Κομισιόν. Ε, τουλάχιστον πολλέ φορέ αναφέρεται η Κομισιόν ως υπεύθυνη. Η Τρόικα στην περίπτωση Ελλάδας και της Πορτογαλίας. Ε, είναι πολύ σημαντικό όταν μιλάμε στην Ευρώπη για διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών αυτές οι αρχές να διέπουν και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ε, η οδηγία πλαίσιο για το νερό που κάνει υποχρεωτική τη διαβούλευση με τους πολίτες στα θέματα διαχείρισης των εντατικών πόρων θα πρέπει να εφαρμόζεται και στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Να έχουν λόγο οι πολίτες και οι φορείς για τα συστήματα διαχείρισης του νερού και τα έργα για το νερό. Όπως επίσης και η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να διασφαλίζει και τους κοινωνικούς όρους, δηλαδή να υποφελούνται αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη, δηλαδή να μην παρέχεται το νερό μέσα από μεγάλα έργα τα οποία αφορούν λίγου, αλλά να φτάνει το πόσιμο νερό και τα αισθήματα αποχέτευσης αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να διασφαλίζει την οικολογική διαχείριση των εντατικών πόρων ε, και να διασφαλίζει ότι προέχει η μη κερδοσκοπική διαχείριση του νερού σε σχέση με άλλε δραστηριότητε. Και τέλο θα πρέπει να διασφαλιστεί και η ε, οικολογική καινοτομία, να υπάρχουν λύσει που είναι κατάλληλε για κάθε περιοχή αλλά και η προστασία των ε, υπόγειων νερών από τη από βιομηχανίες, από εξορίξεις μετάλλων ή χρυσού, εξορίξεις ε, υδρογονανθράκων, σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου στη σχέση μας με άλλες χώρες. Σας ευχαριστώ κύριε Σκυμπράντη για ένα μισό λεπτό. Ναι, συγγνώμη. Άκουγα κάποια άλλη γλώσσα ακόμα. Ναι, συγγνώμη πρόεδρε που καθυστέρησα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εκείνους που συμμετείχαν σε αυτή την πρώτη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Για μένα δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το νερό είναι στο επίκεντρο αυτής της πρώτης πρωτοβουλίας και αυτό γιατί πολύ απλά το νερό είναι ζωή. Και η ζωή είναι το επίκεντρο των όλων των πράξεών μας. Και ασφαλώς είναι ανθρώπινο δικαίωμα το νερό, αυτό είναι προφανές. Αλλά το, να το δηλώνουμε και να το αναγνωρίζουμε αυτό απλά δεν σημαίνει ότι ο κόσμος έχει πρόσβαση στο νερό και στην αποχέτευση. Πολύ πιο σημαντικό είναι, θεωρώ, να εξεταστούν οι όροι και οι συνθήκες οι οποίες θα επιτρέψουν σε μας να εξασφαλίσουμε αυτό το ανθρώπινο δικαίωμα για όλους τον πλανήτη μπορούμε επιμακρών να συζητάμε θέματα απελευθέρωσης ή ε, ιδιωτικοποίησης του νερού, κατά πόσον είναι θετικά αυτά ή όχι, αλλά θα ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο πάροχο του νερού στον πλανήτη, τη φύση. Η φύση η οποία απειλείται με απώλεια βιοποικιλότητας, που απειλεί με τη σειρά τη τη δυνατότητα τη ε, γη να μα παρέχει καθαρό νερό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα καλό παράδειγμα ε, όπου υπάρχει ισχυρή νομοθεσία για την προάσπιση και την προστασία της φύσης. Αυτό το αναγνωρίζω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη δεν το τοποθετούν αυτό απαραίτητα πάντα στην κορυφή του προτεραιότητων Αναγνωρίζω, ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας αναγνωρίζετε ότι η φύση μας παρέχει πάνω απ' όλα το καθαρό νερό και σε ό,τι αφορά τον αγώνα μας θα πρέπει να αγωνιστούμε για την προστασία της φύσης πάνω απ' όλα. Σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye για ένα λεπτό. Λοιπόν, η κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λυπάμαι που έφτασα αρκετά καθυστερημένα πριν από δύο λεπτά, αλλά δυστυχώ είχα συνεδρία σε άλλη επιτροπή. Θα ήθελα να συγχαρώ του οργανωτέ αυτή τη πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών, μια πρωτοβουλία που στέθηκε μεγάλη επιτυχία, πέτυχε το στόχο τη ε, και χαίρομαι και για την ευκαιρία που μα έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη διοργάνωση τη σχετική δημόσια ακρόαση. Είναι σημαντικό λίγου μήνε πριν τι ευρωεκλογέ ε, να λάβουμε υπόψη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας για θέματα τόσο σημαντικά για όλους όπως είναι η πρόσβαση στο είδωρο, στην ίδρυυση και στην αποχέτευση και αναγνώριση αυτών των αγαθών ως θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα πλαίσια της οδηγίας για το νερό υποβάλαμε τις ε, σκέψεις μας και τις διεκδικήσεις μας. Ε, για παράδειγμα την ανάγκη να βρούμε πόρους και στο 1% και όχι μόνο στις ευρωπαϊκές χώρες ε, για να αποφύγουμε να κόβεται το νερό σε άπορες οικογένειες. Θα είπαμε λοιπόν να εξασφαλιστεί πρόσβαση όλων των συμπολιτών μας στο νερό, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες χώρες που δεν έχουν υλοποιήσει ακόμη τους αναπτυξιακούς ε, στόχους της χιλιετίας. Και με βάση την έκθεση ΣΕΒΕΡ ε, ζητήσαμε να χρησιμοποιείτε το 1% των πόρων για να βοηθήσουμε ε, τις άλλες χώρες. Κύριε Επίτροπε Σεφτσοβιτς, ελπίζω να περάσετε σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης, ε, να αναγνωρίσουμε την ιεράρχηση των λύσεων, γιατί σίγουρα είναι το πιο σημαντικό το θέμα των υποδομών. Επίσης, ε, το θέμα της, του διακανονισμού και της επίλυσης διασυνοριακών διαφορών σε θέματα διαχείρισης υδάτων. Αυτό είναι σημαντικό και για την Ευρώπη αλλά και για τρίτες χώρες. Γιατί μερικές φορές ε, το είδωρ γίνεται λόγος για συγκρούσεις. κυρία Παπαδοπούλου, για ένα λεπτό. Και εγώ χαιρετίζω αυτή την πρώτη πρωτοβουλία ε, πολιτών, γιατί είναι η πρώτη ακριβώ που συγκέντρωσε 2 εκατομμύρια υπογραφέ μετά την εφαρμογή τη ηθίκη τη Λισαβόνα. Και είμαι σίγουρη, γιατί ήμουν η συγγραφέα τη έκθεση για το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτών, πρέπει να αναπτύξουμε τη συμμετοχική δημοκρατία και την ενεργό πολιτότητα. Και έχει πολλά που μπορούμε να κάνουμε για του Ευρωπαίου πολίτε και όχι μόνο. Ε, αυτό το οποίο εμένα με ξενίζει είναι η μεγάλη ανισότητα που υπάρχει όσον αφορά τη χρήση του νερού. Στην Ευρώπη υπάρχει οδηγία πλαίσιων, υπάρχουν αυστηρέ προδιαγραφέ. Προσωπικά ήμουν για 23 χρόνια διευθυντή ελέγχου ποιότητα και ήμουν υπεύθυνη για το χημικό μικροβιολογικό έλεγχο του νερού. Και είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούνται αυτέ οι οδηγίε. Όμως σε πολλές χώρες, στην Αφρική, στην Ασία, αυτές οι οδηγίες δεν ακολουθούνται. Και εδώ υπάρχει μια τεράστια ανισότητα. Εκείνο όμως που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η Τρόικα στις χώρες του Μνημονίου. Δυστυχώς, όπως έχει πει και ο συνάδελφος από την Ελλάδα, ο κύριος Χρυσόγελος, ιδιωτικοποιεί διάφορα αγαθά. Και αυτό που με ξενίζει είναι με τις ιδιωτικοποιήσεις αν τελικά το νερό θα πάψει να είναι ανθρώπινο δικαίωμα και σε αυτήν ακόμα την Ευρώπη και το κέρδος, η εσχροκέρδεια κυρίω, θα πριτανεύσει γιατί ζούμε σε μια εποχή κρίσης αξιών και αυτό είναι κάτι που με φοβίζει ιδιαίτερα. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, γιατί ο κύριος Ρεν λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Τηρεί στα ουδέτερη. Τότε ποιο επιβάλλει αυτή ε, τη δράση της Τρόικας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι γίνεται. Σας ευχαριστώ ο κύριος Χέφνερ για ένα μισή λεπτό. Ναι, αυτό που με απασχολεί εδώ και μιλώ τώρα και από πλευράς της Επιτροπής Αναφορών είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά με τη ECI, με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία, αναπτύξαμε ένα είδος ε, γλώσσας ε, για τους πολίτες. Μας ε, φέρνετε αντιμέτωπους και αυτό ισχύει και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μια πολύ βασική συζήτηση σε ό,τι αφορά τη μακροπρόθεσμη ε, το μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της πολιτικής μου και προσπαθώ λοιπόν να σκεφτώ πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο. Ένα παράδειγμα να σας δώσω εδώ. Έχουμε λοιπόν 1,9 ε, ε, εκατομμύρια πολίτες που τάσσονται κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού και υπάρχει λοιπόν αυτή η τάση, αυτή η πλειοψηφία του κόσμου στην Ευρώπη που τοποθετείται έτσι, ιδιαίτερως και στις χώρες εκείνες που έχουν γίνει μαζικώς ε, ιδιωτικοποίησης, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι η Τρόικα ως ευρωπαϊκός θεσμός στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, επιβάλλει ιδιωτικοποίηση του νερού. Ερωτώ λοιπόν τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι η πολιτική αυτή που επιθυμούν οι πολίτες οι Ευρωπαίοι θα είναι η πολιτική που θα ασκεί η Τρόικα. Πώς μπορούμε στην πολιτική, την εξωτερική, στην ε, αναπτυξιακή συνεργασία, να διασφαλίσουμε ότι αυτό το απίστευτα σημαντικό θέμα για όλους τον πλανήτη θα το αντιμετωπίσουμε με τέτοιο τρόπο προκειμένου να μην είναι μελλοντική πόλεμη για το νερό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κοινό καθεστώς, χρειαζόμαστε κοινά αποδεκτούς διεθνείς κανόνες. Πώς θα τα πετύχουμε αυτά και πώς θα πετύχουμε αυτό να το προασπίσουμε και στην εξωτερική πολιτική. Αυτό που θέλει ο κόσμος, όχι αυτό που θέλουν οι ιδιωτικοί όμιλοι και τα συμφέροντά τους. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κύριε Χέφνερ και τώρα το λόγο έχει η Επιτροπή των Πολιτών για 10 λεπτά για να απαντήσει στις ερωτήσεις που ακούσαμε. Σας παρακαλώ να αποφασίσετε εσείς σε ποιον θέλετε να βάσετε το λόγο, αλλά 10 λεπτά αυτό είναι το χρονοδιάγραμμά μας. Ε, Ευχαριστώ ξεκινώ εγώ και ίσως μετά δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Έχω την αίσθηση, καταρχάς να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω που θέσατε ένα τόσο ε, σημαντικό ερώτημα. Πώς δηλαδή προστατεύοντας και επιβεβαιώνοντας το δικαίωμα πρόσβαση στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα, ε, θα μπορέσουμε να προβλέψουμε και τις διαδικασίες ώστε αυτό το δικαίωμα να προστατεύεται στην πράξη. Πιστεύω ότι το να προστατεύουμε ένα ανθρωπίνο δικαίωμα σημαίνει ότι θα λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν μπορεί να είναι εμπορεύσιμο αγαθό το νερό ή τουλάχιστον ένα αγαθό επί του οποίου διοργανώνονται εμπορικές δραστηριότητες με σκοπό την αποκόμιση κέρδους. Υπάρχουν και κάποια δεδομένα για να καταλάβουμε πώς έχει κατάσταση. Τα τελευταία 10 χρόνια, από το 2001 και τα τελευταία 13 συγκεκριμένα χρόνια, βιώνουμε μία επιστροφή στις πολιτικές ιδιωτικοποίησεις για τις υπηρεσίες του νερού. Στις τελευταίες 86 υποθέσεις που λάβαμε υπόψη από αυτές, 51 ε, συνέβησαν σε χώρες με υψηλό εισόδημα εκ και 35 σε αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες έλαβαν χώρο στη Γαλλία που ξέρετε ότι έχει περάσει στα χέρια των μεγάλων πολυεθνικών του νερού. Έτσι το Παρίσι ως πόλη και ως Δήμος έλαβε την απόφαση να ξαναπάρει στα χέρια του τη διαχείριση του νερού. Αυτέ είναι διαδικασίε που αναλαμβάνονται και σε πολλέ άλλε χώρε, 15 μεγάλε πόλεις στι ΗΠΑ που είχαν ιδιωτικοποιήσει το νερό έδωσαν τέρμα στη σύμβαση αυτό τη σύμβαση αυτή για την ίδρυυση και από τι 15 αυτέ τι πόλει. 12 είχαν αναθέσει την ίδρυυση σε μεγάλες πολυεθνικές της Ευρώπης. Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, όπως την ανάκτηση της ίδρυυτη της Λαπάς, του Μπενοσάιρας, του Γιωχάνεσμπουργκ, του Νταραλ Σαλάμ, στην Κάνα και η συζήτηση ξαναρχίζει για το θέμα αυτό και στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι στον κόσμο όλοι διερωτώνται για την ποιότητα της υπηρεσίας που μπορεί να προσφέρουν οι ιδιωτικέ εταιρείε. Και η απάντηση που ως επιτοπλίστων δίνεται είναι ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί περισσότερο να διασφαλίσει το δικαίωμα αυτό ανθρώπινο, την πρόσβαση στο καθαρό νερό και την παροχή της υπηρεσίας με χαμηλό κόστος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληρώσουν αυτό το αγαθό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι περιορίζεται το κέρδος μιας ιδιωτικής εταιρείας. Δεν είναι το ίδιο ένας δημόσιος φορέας. Και αυτό συμβαίνει σε χώρες τελείως διαφορετικές μεταξύ τους με χώρες τελείως διαφορετικής ε, προέλευσης και μπορεί να κυβερνώνται από τελείω διαφορετικού συνασπισμού ή πολιτικέ πραγματικότητε. Αυτό που ζητάμε εμεί ω πολίτε, ω Επιτροπή των Πολιτών, είναι ότι εμείς πιστεύουμε ότι δεν αρκεί μία επί της αρχής επιβεβαίωση προστασία του δικαιώματος αυτού. Έχουμε πάρα πολλές μαρτυρίες και αποδείξεις γι' αυτό. Θέλουμε συγκεκριμένους δείκτες, κριτήρια που να λαμβάνουν υπόψη τον σεβασμό αυτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις πολιτικές που εκπονεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει και το θέμα αυτό το έθιξαν και οι εκπρόσωποι της Ισπανίας, της Ελλάδας, θα ήταν ωραίο να πει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τρόικα, αποκλείει από τις ιδιωτικοποίησεις την διαχείριση του νερού, την ίδρυψη της Θεσσαλονίκη εφόσον ε, υλοποιούνται εκεί ε, πολιτικές λιτότητας. Εφόσον είναι ανθρώπινο αγαθό το νερό να παραμείνει στα χέρια του Δήμου, ε, ε, του δημόσιου τομέα. Επίσης να τονίσω ότι για κάθε δολάριο που επενδύουμε στον τομέα αυτό έχουμε επιστροφή του, της σε πολύ μεγάλο ποσοστό και ως προς την κερδοφορία της επένδυσης της ίδιας και την κερδοφορία γενικότερα για την ε, κοινότητα την κοινωνία, διότι προσδίδει μεγάλα κοινωνικά ωφέλη, μικρότερο κόστος για την υγεία των πολιτών, μικρότερο κόστος για την περίθαλψή τους, για την προστασία του περιβάλλοντος, διότι ακριβώς ο δημόσιος τομέας ε, προστατεύει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά την, ε, το αποθεματικό αυτού του φυσικού πόρου και το πώς διοχετεύεται ή όχι στην φύση. Και κάτι άλλο, στις ευρωπαϊκές πολιτικές έχει υποτιμηθεί αυτό το στοιχείο, αλλά γίνεται μια κατεπίγουσα ανάγκη παγκοσμίω. Να πω ότι συμμετέχω και στον ΟΗΕ, στην ομάδα, το Συμβουλευτικό Φόρουμ ε, της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά και προσφάτως συζητήσαμε το θέμα αυτό και οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών εταιριών μας είπαν ότι όχι, όχι, είμαστε πανέτοιμοι να ικανοποιήσουμε την ανάγκη των πολιτών, ιδίως αν υπάρξουν και καταστροφές που έχουν σχέση με το νερό. Μπορούμε να παρέμβουμε, αλλά μόνον αφού έχουν επανέλθει οι συνθήκες πρόσβαση στην υπηρεσία. Ιδού, ο δημόσιος τομέας όμως λαμβάνει δράση ακόμη και όταν υπάρξουν ε, κατεπίγουσες ανάγκες σε καταστροφές που έχουν σχέση με την πρόσβαση στο νερό και φροντίζει να αποκατασταθεί η παροχή της υπηρεσίας και όλη τη συνέχεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα έπρεπε να προβλέψει σχέσεις συνεργασίας, πολιτικής συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες ή τουλάχιστον στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών να λαμβάνεται υπόψη και αυτός ο παράγων. Δηλαδή ότι όταν μιλάμε για νερό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι διασφαλίζουμε ένα ανθρώπινο δικαίωμα και πρόσβαση στο νερό και στις υπηρεσίες ε, αποχέτευσης, προστασίας ενός φυσικού πόρου γενικότερα και αποφεύγουμε να γίνει ένα όχημα ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αυτού αγαθού σε πολλέ χώρε, διότι οι μορφέ ιδιωτικοποίηση, όπω είδαμε, μπορεί να είναι συντεκαλυμμένε. Απελευθέρωση ιδιωτικοποίηση μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν, αν εγγυηθούμε την πρόσβαση στον, στους πολίτες στο νερό με χαμηλό κόστος, είναι ήδη σημαντικό αυτό και πρέπει να αναπτύξουμε πολιτικές που να επιτρέπουν τη συνεργασία του δημόσιου με τον δημόσιο φορέα, δηλαδή συνεργασία των δημόσιων φορέων της Ευρώπης μεταξύ τους. Υπάρχουν και είναι πολύ σημαντική. Και είναι σημαντική και για την ανατόνωση των τοπικών οικονομιών. Και έτσι μπορεί να ευνοηθεί η οικονομική ανάπτυξη και σε τρίτες χώρες κατ' επέκταση σε εξωευρωπαϊκές χώρες, δεδομένων των τοπικών συνθήκων, δεδομένης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας εκεί, δεδομένης της ανάπτυξης που όπως μας δείχνει η κρίση δεν μπορεί πλέον να υπόκειται μόνο στην ε, ρύθμιση της απαιτήσει της παγκοσμιοποίησης όπως έχει διαμορφωθεί ως σήμερα. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να ανταποκριθεί με ικανοποιητικό τρόπο τι διεκδικήσει, τι απαιτήσει και τι εκκλήσει τη ε, Οργανωτική Επιτροπή τη ε, Πρωτοβουλία των Πολιτών. Αλλά καταρχά θα έπρεπε να ακούσει, να ακούσει η Ευρώπη το λαό τη. Αυτό θα απεδείκνυε το να ληφθούν υπόψη ε, οι απαιτήσει μα, να πάψει αυτή η καχυποψία που έχει δημιουργηθεί και ο να γίνουμε ένα μοντέλο για τον υπόλοιπο κόσμο, για την προστασία των κοινωνικών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Νομίζω ότι υπάρχει λίγος χρόνος ακόμα, 1,5 λεπτό. Στο 1,5 λεπτό που έχει απομείνει, θα ήθελα να πω στον Τζάραλ Χέφνερ ότι βέβαια το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό στον κόσμο δεν θα υλοποιηθεί αν δεν δώσουμε μάχη για να ανακτήσουμε την... και να αποκαταστήσουμε τα υδάτινα οικοσυστήματά μας και τον υδρολογικό κύκλο. Γιατί τα... και οι φτωχοί χρειάζονται καθαρά ποτάμια. Δεν είναι μόνο πρόβλημα των πλούσιων και των ευπόρων. Αλλά οι φτωχοί και οι άποροι είναι αυτοί που ξεκινάν τον αγώνα κατά της ε, καταστροφής ε, του, του, των πολιτών. Και Νίκο, τα ορυχεία σε όλη τη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, ε, δημιουργούν τοξικά απόβλητα και τα αγροτοξικά στοιχεία ενισχύουν την τοξική ρήπανση που βάζουμε στους σωλήνες και μάλιστα με εκθετικό τρόπο. Και δεν έχουμε καν διεθνούς υπολογισμούς. Οι 10.000 θάνατοι καθημερινά είναι από διάρειες, από βιολογική ρήπαση και στη Λίμα... Ε, στην τελευταία συνάντηση που είχα με τα συνδικάτα μου είπαν στη Λίμα 9 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν δικαίωμα σε πόσιμο νερό γιατί το πολύ το, ποτάμι ε, έχει μολυνθεί από βαριά μέταλλα εξαιτίας της εξορυκτικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν πώς παράγουμε τις, ε, τους σπόρους. Αγροτοξικά στοιχεία, φράκινγκ, ε, υδρορογμάτωση. Θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο γίνεται και αυτή η παραγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Κλάουζ Ρούντι Σάουζερ. Τέσσερα λεπτά έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρίε και κύριοι να πω ότι είναι τιμή μου και χαρά μου που συμμετέχω εδώ σήμερα στη συζήτηση αυτή και πιστεύω ότι έχουμε πραγματικά κάποια πράγματα να συμβάλλουμε στη συζήτηση αυτή. Η... Το νερό και η αποχέτευση ήταν και θα είναι πάντα ένα κεντρικό θέμα της αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό περιλαμβάνεται και ε, σε όλα τα έγγραφα τα σχετικά και νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο παρέχει 60% της αναπτυξιακής βοήθειας, είναι ένας από τους προδρόμους αυτής της υποστήριξης της πρωτοβουλίας αυτής δεν νομίζω ότι υπερβάλλουμε. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να το πούμε αυτό. Και ιδιαίτερος επειδή πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, το οποία εμείς ξοδεύουμε σε τρίτες χώρες και έτσι λοιπόν μεταφέρουμε τα συμφέροντά σας σε τρίτες χώρες. Κάποια παραδείγματα μόνο. Δεσμευτήκαμε στην επόμενη πραγματική περίοδο να δώσουμε 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τον υποσυτισμό και επειδή ο υποσυτισμός συχνά έχει να κάνει και με τα θέματα υδροδότησης και αποχέτευσης και όχι τόσο με θέματα τροφίμων, σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα των κονδυλίων αυτό θα δαπανηθεί για την ε, επεξεργασία λιμάτων και για την υδροδότηση. Στην ε, τρέχουσα περίοδο μέχρι το 2013 επενδύσαμε 2,3 δισεκατομμύρια μόνο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό σε, σε αναπτυξόμενες χώρες, σε χώρες τέτοιες εταιρικής σχέσεις και ένα μεγάλο τμήμα των κονδυλίων αυτών. Πιστώσεις σε ύψος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν δοθεί, έχουμε υποστηρίξει δηλαδή τέτοιες πιστώσεις σε αναπτυξιακές τράπεζες. Άρα είναι πολύ πιο μεγάλο το ποσό αυτό αν προσθεθούν και οι πιστώσεις. Λοιπόν, τίθεται ένα θέμα δικαίου. Φυσικά η πολιτική αναπτυξιακή μας βασίζεται σε όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, σε όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ και άρα δεν τίθεται καν το ερώτημα. Αν δεσμευόμαστε για το θέμα του νερού, Βασιζόμαστε λοιπόν στις νομικές αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ζήτηση. Να επικεντρώσουμε δηλαδή τα κονδύλια μας εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η σημασία του νερού αναγνωρίζεται, το επισήμανε αυτό και η κυρία Στρίφλερ, πρόκειται για ένα από τους στόχους της χιλιετίας και πρόκειται για έναν στόχο τον οποίο, στον οποίο υπάρχει όντως μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν το νερό θα συνεχίσει να παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας, αλλά αυτό που είναι ακόμα πιο ουσιώδες είναι στο μέλλον να ορίσουμε με καλύτερο τρόπο και διάφοροι ομιλητέ το έθιξαν αυτό. Σε 1,5 χρόνο στη Νέα Υόρκη θα υπάρξει μια νέα αναπτυξιακή ατζέντα για την περίοδο μετά το 2015 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις τρέχουσες ανακοινώσεις της για το θέμα αυτό ή την προσοχή στην ε, υπεύθυνη αντιμετώπιση και χρήση των φυσικών πόρων. Αυτό τι σημαίνει ότι στη Νέα Υόρκη λοιπόν θα ταχθούμε υπέρ της ε, γραπτής συμπερίληψης αυτής της υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων. Να μπει αυτό στο κείμενο. Κάποια άλλα σημεία τα οποία θεωρώ είναι σημαντικά και τα οποία θα έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη. Καταρχάς είπαμε ότι υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό τι σημαίνει ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάποια χώρα κάνει κάτι λιγότερο στο θέμα του νερού, κατά κανόνα δραστηριοποιούνται κράτη-μέλη, ένα ή περισσότερα ή κάποιες οργανώσεις στη χώρα αυτή. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτή η κατανομή των εργασιών. Και τι άλλο όμως είναι σημαντικό, η συνεργασία, η αναπτυξιακή πρέπει πάντα να είναι βοήθεια για αυτοβοήθεια. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Χρειαζόμαστε και τη συμμετοχή των κυβερνήσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αυτό είναι μια σημαντική πρόκληση σε διπλωματικό επίπεδο για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή την, αυτό το καθήκον το έχουμε υπόψη μας θα ήθελα να επαναλάβω χωρίς να επισέλθω σε υπερβολικές λεπτομέρειες ότι ο στόχο τη πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο της αναπτυξιακή μα συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρο και τώρα το λόγο έχει, έχει κλείνοντας η κυρία Παβανέλη. Έχετε το λόγο λοιπόν για να κλείσετε και αυτό το γύρο ερωταπαντήσεων. Ε, ε, ναι, πολύ σύντομα νομίζω είναι σημαντικό στις αναπτυξιακές μας πολιτικές όλο και περισσότερο να λαμβάνουμε υπόψη του γεγονότος του ότι το νερό είναι σημαντικό όχι μόνο για να εξασφαλίσουμε κάθε μορφή ζωής, ακόμη και την ανθρώπινη, αλλά ότι ως ε, στοιχείο σχετίζεται όλο και περισσότερο με τις ενεργειακές μας πολιτικές και τις πολιτικές επισητιστικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό το να επιβεβαιώσουμε ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα είναι στοιχείο που είναι απαραίτητο ε, τη στιγμή που μιλάμε για τις επιστημιστικές προοπτικές ενός πλανήτη του οποίο ο πληθυσμό αυξάνεται και σύντομα μπορεί να μην υπάρχουν αρκετά τρόφιμα για να μπορούν όλοι να τραφούν και να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Από αυτήν τη σκοπιά ένα στοιχείο μου φαίνεται πολύ σημαντικό και πρέπει να τονιστεί. Δηλαδή, αφού αναγνωρίζουμε ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα, θα πρέπει να αποκλειστεί όχι μόνο από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς, αλλά και από τις διαπραγματεύσεις ελεύθερων συναλλαγών, απελευθέρωσης του εμπορίου που έχουμε σε πολλές μορφές με τις ε, σχέσεις, τις συμφωνίες συνεργασίας, τις ε, τρικες σχέσεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες όπως είδατε έχουν ασκήσει την πρωτοβουλία τους, ασκούν πίεση και ελπίζουμε ότι το την πρωτοβουλία θα συνεχίσουμε με θετικό τρόπο στην ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, και έτσι λοιπόν ολοκληρώσαμε και το δεύτερο γύρο. Να αλλάξουμε και πάλι σύνθεση και να συνεχίσουμε μετά με, τρίτο, με την τρίτη ενότητα, όχι στην απελευθέρωση των ε, υπηρεσιών υδροδότησης. Να αλλάξουμε λοιπόν τα έδρανα και να προετοιμαστούν οι επόμενοι ομιλητές. So, ich bitte doch alle, die Plätze wieder ein. Σας παρακαλώ καθίστε λοιπόν στις θέσεις σας για να ξεκινήσουμε λοιπόν και με τον τρίτο γύρο, την τρίτη ενότητα. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ότ για πέντε λεπτά. Θα μας παρουσιάσει τους στόχους. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γκρότα. Στη συζήτηση πολλά ακούσαμε ήδη. Εμείς, ε, ποια είναι η επικεφαλή μας, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα πάνω από τα συμφέροντα της αγοράς. Όχι στην απελευθέρωση λοιπόν των ε, ε, οδηγιών των ε, υπηρεσιών για την υδροδότηση. Αυτό είναι φυσικά κάτι που γνωρίζουν όλοι. Πρόκειται για ένα κοινοφερέ αγαθό το οποίο είναι ύψη τη σημασία για την ασφάλεια και τη ζωή. Η πρόσβαση λοιπόν στην ε, υδροδότηση και στην αποχέτευση είναι προπόθεση για άλλε βασικά θεμελιώδη δικαιώματα όπω η υγεία ή για την παιδεία για παράδειγμα. Και γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζουμε ότι δεν είναι αγαθό το νερό. Λέγοντα ότι το νερό δεν είναι αγαθό, τι θα πρέπει να διασπαθεί να διαπιστώσουμε ποιος είναι αυτός ε, που εμπορεύεται τα αγαθά. Οι ιδιωτικές εταιρείε. η δουλειά τους και η στοχοθέτησή τους όμως δεν είναι να εκπληρώσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι απλά πρέπει να τα τηρούν. Ποιοι θα πρέπει να επιβάλλουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος καταρχάς. Αυτό τι σημαίνει ανθρώπινο δικαίωμα είναι και η διασφάλιση της πρόσβασης στο νερό. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία θα πρέπει να διοργανωθεί όσο πιο κοντά γίνεται στον πολίτη και ο δημοκρατικός ε, έλεγχος και η συμμετοχή η δημοκρατική αυτή του πολίτη θα πρέπει να διασφαλίζεται. Και αυτό λοιπόν ε, σημαίνει ότι έχουμε ιδιαίτερα καθήκοντα. Το νερό αποτελεί ένα φυσικό μονοπόλιο και δεν θα πρέπει σε αυτό να εφαρμοστούν οι κανόνες της ε, ενιαίας κοινής αγοράς οι δήμοι και οι κοινότητες θα πρέπει να είναι πάσα στιγμή υπεύθυνε και να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό γιατί είναι μια δημοκρατική, μια δημοκρατική αρχή και η αρχή του δημοκρατικού ελέγχου επιβεβαιώνεται έτσι. Γι' αυτό λοιπόν τη ζητούμε το νερό και οι υδάτινοι πόροι να ανακηρυχθούν δημόσιο αγαθό και η εμπορία, μάλλον η διαχείριση του, των υδάτινων πόρων να μην υπόκειται στους κανόνες της αγοράς. Ένα ψήφισμα δεκαετές πλέον. Το 2004 το αποφάσισε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ανέκρινε. Αυτό τι σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το νερό για κέρδος. Όλοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο νερό και αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί με σαφέστατο τρόπο στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Καλωσορίζουμε το γεγονός αυτό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτέλεσε το βασικό στόχο της πρωτοβουλίας, το γεγονός ότι το νερό εξαιρέθηκε από την οδηγία παραχώρησης. Προκειμένου λοιπόν το νερό να αφαιρεθεί από την οδηγία παραχώρησης και έτσι να διευκρινιστεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο το δικαίωμα στην υδροδότηση. Τι άλλο. Υπάρχουν ε, σημαντικές ε, αμφιβολίες και ανησυχίες κατά της συμπερίληψης της ε, υδροδότησης, της διαπραγματεύσεις για ζώνες ελευθέρου εμπορίου, όπως τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται σήμερα με, την, με τη ΣΥΠΑ. Γιατί αυτό αντιτίθεται στις αρχές της ελεύθερης πρόσβασης στο νερό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες εταίρους με τις οποίες διεξάγονται διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν οι διαδικασίες διαμεσολάβησης ενδεχομένως να έχουν και ένα μη υπολογιζόμενο κόστος για τους Δήμους και τις κοινότητες σε ό,τι αφορά α, την υδροδότηση και την Αποχέτευση. Ενδεχομένω δηλαδή να υπάρχει και υπερβολικό αριθμό καταγγελιών σε περίπτωση απελευθέρωση του κλάδου αυτού. Έχουν θεθεί, τέτοια ε, benchmarks και σε εθνικό επίπεδο εδώ και πάρα πολύ καιρό και στην Γερμανία για παράδειγμα και στην Ολλανδία και ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας και η βελτίωση της ασφάλειας σε ό,τι αφορά την ευρωδότηση. Αυτός είναι ο στόχος δεδομένων του, του υψηλού κόστου σε ό,τι αφορά την ενδρότηση, βασικό είναι να χρησιμοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια και να διδασκόμαστε από τις ε, βέλτιστε εμπειρίε των άλλων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδράμει και το δικό τη ε, από, το, από δική της πλευράς. Κάτι άλλο τώρα σε ό,τι αφορά τους Δήμους της Κοινότητας και τις ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις τροδοζώτησης. Όσοι δήμοι και κοινότητες ε, αποδέχονται την ιδιωτικοποίηση, ουσιαστικά αποδέχονται την κερδοσκοπία σε ό,τι αφορά αυτό το φυσικό αγαθό. Αν ο δημοκρατικός έλεγχος ε, δεν υπάρξει και δεν είναι επαρκής, θα πρέπει να υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις τροφοζώτησης θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται τα κέρδη και οι πολιτές και οι εκπρόσωποι του στου Δήμου και τι κοινότητε θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην απόφαση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευρωπαϊκού κανόνε για τη συμμετοχή, τη διαφάνεια. Και σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Θα πρέπει να προσέξουμε το χρόνο γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις 6.30 μόνο γιατί μετά οι διερμηνεί θα αναγκαστούν να φύγουν. Γι' αυτό λοιπόν να ζητήσω από όλους τους ομιλητές να είναι σύντομοι, να τηρήσουν το χρονικό όριο που τους δίδεται. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν ε, το γύρο των ερωταπαντήσεων. 1,5 λεπτό στον κάθε ε, ομιλητή. Λεκή. 1,5 λεπτό παρακαλώ, η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω εισαγωγικά ότι κατά τη γνώμη μου το θέμα της πρόσβασης στο νερό δεν είναι θέμα ιδεολογίας. Είναι θέμα δικαίου ή δικαιώματος, προτεραιότητας, δράσης και αποτελεσματικότητας. Πώς να διαφωνήσουμε με τα σημεία 1 και 3 της πρώτης αυτής της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών. Προφανώς και συμφωνούμε και ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συμφωνώ με το αίτημα της δεύτερης παραγράφου που λέει ότι η υδροδότηση δεν θα πρέπει να εμπίπτει στους κανόνες της εσωτερικής αγοράς και να αποκλείεται από την απελευθέρωση. Το σημείο 2 βέβαια είναι κάπως αμφίσιμο ε, ίσως είναι σκεμμένη αυτή η σύγχυση μεταξύ του ύδατος αφενός και των συναφών υπηρεσιών αφετέρου. Γιατί στο παράρτημα ή στο επεξηγηματικό σημείωμα που είναι πολύ εντελεχές και που περιλαμβάνει ένα κατάλογο με 10 προτάσεις από την Επιτροπή της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων Πολιτών αναφέρεται ότι μόνο το είδωρος, φυσικός πόρος θα πρέπει να αποκλείεται από τους κανόνες εσωτερική εσωτερικής αγοράς. Λοιπόν, γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση στην παράγραφο 2 και γιατί αυτή η αφησιμία. Το είδωρ είναι ένα αγαθό, ένα δικαίωμα, ένας φυσικός πόρος που θα πρέπει να τύχει δικής προστασίας και η σχετική οι συναφεί υπηρεσίε και οι υπηρεσίες διαχείρισης υδροδότησης θα πρέπει και αυτέ να αποκλείονται από την εσωτερική αγορά. Θα ήθελα όμω να διευκρινίσετε. Επίση, να υπενθυμίσω ότι οι τη εσωτερική αγορά που ισχύουν και για τι υπηρεσίε ε, γενικού συμφέροντο και άρα και των υπηρεσιών νερού εξασφαλίζουν μια διαφάνεια, ισότητα μεταχείρισης, αποφυγή τη διακριτική μεταχείρισης μεταξύ χρηστών και παρόχων στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε υπόψη το συγκεκριμένο συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, από πιθανά μέτρα που θα θεσπίσει στο μέλλον, το απότερο μάλλον μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά την τιμή, την προσπελασιμότητα και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων και των μελλοντικών υποδομών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Γκέπχαρτ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Ότε. Σωστά μόλις υποδείξατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση του νερού ως ενός γενικού αγαθού για όλους τους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το νερό να γίνει έρμενο, έρμεο του προσανατολισμού και των συμφερόντων της ε, αγοράς. Και κάτι άλλο που αναφέρατε, τις ε, συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης, όπου υπάρχει και ένα κεφάλαιο για τις δημόσιες προμήθειες και για τις υπηρεσίες γενικού κοινοφιλούς ε, συμφέροντος. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να μας πει πώς τοποθετήσετε σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Αυτή την έκκληση των 1,9 εκατομμυρίων πολιτών και πολλών ακόμα που δεν υπέγραψαν κατά πάσα πιθανότητα, πώς θα φροντίσετε να μην καταλήξουν όλοι οι καλοί κανόνες που καταρτίζουμε εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διακυβεύονται πολύ απλά επειδή υπάρχει μια προστασία επενδύσεων. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Υποδειγματική λοιπόν η Εύελιν Γκέπχαρτ τήρησε το των 1,5 λεπτών η πρώτη ομιλητρία που το κατάφερε. Μάλιστα. 1,5 λεπτό η συνάδελφο ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Πρωτοβουλία των Πολιτών και σκεπτόμενοι το πώς συζητήσαμε τα θέματα παραχωρήσεων ε, ε, υπηρεσιών παραχώρησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα καταφέραμε να τις εξαιρέσουμε να το νερό από τις συμβάσεις παραχώρησης και, φυσικό, φυσικά δεν πρόκειται για την ε, ιδιωτικοποίηση, για τα θέματα Αυτά είναι θέματα των ε, κρατών μελών. Το θέμα είναι η απελευθέρωση. Και γι' αυτό λοιπόν το νερό ευτυχώς εξαιρέθηκε από τις συμβάσεις παραχώρησης. Χαίρομαι λοιπόν που το νερό δεν θα υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες για την απελευθέρωση. Δεν ήταν η πρώτη της τέτοιος αγώνας. Χαίρομαι που τον κερδίσαμε. Αλλά, αλλά το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εξής. Αυτό το πετύχαμε μόνο μέσω ενός συμβιβασμού. Ο συμβασμός αυτός τι έλεγε, ότι θα υπάρχει μια ρήτρα αναθεώρηση. Σε δύο συν τρία χρόνια λοιπόν θα ελεγχθεί κατά πόσο, ποιος είναι, είναι ο αντίκτυπος αυτής της εξέριξης του νερού. Όχι ποιος είναι ο αντίκτυπος στην ενιαία αγορά, αυτό το αποφύγαμε. Ποιος είναι ο αντίκτυπος λαμβάνοντας υπόψη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του νερού. Ρωτώ λοιπόν αυτό. Πώς θέλετε να το κατήσετε, πώς θέλετε να το ορίσετε επακριβώς και να ερωτήσω και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία. Τι ζητάτε, τι απαιτείτε. Πρόκειται για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν θέλουμε σε πέντε χρόνια η μοναδική επιτυχία που σημειώσαμε να αναιρεθεί. Τι θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε. Πολύ συγκεκριμένα και θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε εκ νέου ότι το νερό δεν είναι ένα συνηθισμένο αγαθό, αλλά και ότι οι υπηρεσίε που έχουν να κάνουν με το νερό δεν μπορούν να είναι ανοιχτέ σε απελευθέρωση και σε δυτικοποίηση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ρούλε. Δεν είστε γιόγκ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενάμιση, ενάμιση διορθώνει ο πρόεδρο, Ενάμιση λεπτό. Φρίκι στα πρόσωπα των συναδέλφων είδα. Όχι, ενάμιση λεπτό μόνο έχετε. Ναι, και εγώ που νόμιζα ότι είσαστε τόσο καλο μαζί μου, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του υπεύθυνου για την πρωτοβουλία αυτή. Στην Επιτροπή Ιστορικής αγορά. Ε, προσπαθούμε να πετύχουμε την καλή λειτουργία τη ε, ιστορικής αγορά, αλλά θα πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν και όρια σε ό,τι αφορά την ιστορική αγορά, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, σε ό,τι αφορά τι κοινοφιλεί υπηρεσίε. Ε, Δηλαδή, συμφωνώ για την εξαίρεση από τις συμβάσεις παραχώρησης, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσω και με την κυρία Ρούλε ότι θα πρέπει να ζητήσουμε εξασφάλιση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν θα αλλάξει αυτό στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προφανώς εξακολουθεί να υποστηρίζει την ιδιωτικοποίηση. Δάλλας δεν θα το υποστηρίζει αυτό στις χώρες εκείνες. Πώς μπορείτε λοιπόν να δείχνετε τέτοια ανισορροπία, να συμφωνείτε σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις της παραχώρησης, αλλά να συμφωνείτε και με την Τρόικα. Δύο προκλήσεις βλέπω για το μέλλον. Καταρχάς στην Ολλανδία βλέπω ότι οι επιχειρήσεις υδροδότησης έχουν κίνητρα στο εξωτερικό να λειτουργήσουν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ στο ιστορικό της χώρας από το πράττουν αυτό. Είναι κοινοφελείς υπηρεσίες, ποια η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια η άποψη και της πρωτοβουλίας, δεν είναι επικίνδυνο αυτό και να συμφωνήσω με τις ερωτήσεις που έθεσε και η Ευελίνη Κέπχαρτ σε ό,τι αφορά τη συνθήκη με την Αμερική. Αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα ήθελε να επανέλθει ε, η υδροδότηση στα δημοσία χέρια, δεν θα έχει προβλήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επιτροπή των Πολιτών για να απαντήσει στα ερωτήματα που ετέθησαν. Οκτώ λεπτά. Ähm, Θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που έχουν να κάνουν με τη σχέση μεταξύ της πρωτοβουλίας και τη... των εκκλήσεών σας σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης. Είπα προηγουμένως ότι οι συμβάσεις παραχώρησης δεν ήταν στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας. Αυτό το είπα λοιπόν προηγουμένως. Αλλά στη δημόσια συζήτηση υπησύλθε με διαφορετικό τρόπο από ότι κατά το παρελθόν σε ευρωπαϊκό προσκήνιο. Χαιρόμαστε λοιπόν το, για το γεγονός που εξαιρέθηκε ο τομέας του νερού. Αλλά βλέπουμε και το παραθυράκι μέσα από τα ρήτρα αναθεώρησης, η οποία ε, στο αποτέλεσμα, τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει, άνοιγμα της αγοράς ε, και συμπερίληψη του θέματος του νερού. Να τεθεί αυτό εκ νέου στην ημερήσια διάταξη. Άρα είναι απαραίτητο να το εξετάσουμε αυτό από πλευρά τη πρωτοβουλία και να πούμε ότι αναγνωρίζουμε ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν άνοιγμα τη ιστορική αγορά. και αυτό το εξασφαλίζουμε, το εγγυόμαστε για το μέλλον. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από το να λέμε ότι θέλουμε να υπάρχει ε, υποστήριξη του ανθρώπινου δικαιώματος για το νερό. Όχι, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό καθήκον και αυτό έχει να κάνει και με τις υπηρεσίες συντροτότητας και όχι μόνο με το αν είναι εμπόρευμα και αγαθό το νερό ή όχι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να απαντήσω στην κυρία Λεγκρίπ, την ε, Ευρωβουλευτή από τη Γαλλία, που φαίνεται ότι είναι υπέρ των στόχων 1 και 3 της πρωτοβουλίας για την πρόθεση του νερού ως ανθρώπινου δικαιώματος και την συμπερίληψή του στις ε, πολιτικές ένωσης, αλλά είστε υπέρ και της απελευθέρωσης και το κόμμα σας υπέρ της απελευθέρωσης των υπηρεσιών νερού. Όχι, εμείς αυτό ζητήσαμε, τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην απελευθερώσει τις υπηρεσίες υδροδότησης. Θέλουμε μια δεσμευτική και υποχρεωτική ανάληψη, ή πρόταση νομοθετική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη απελευθέρωση των υδροδοτικών υπηρεσιών. Και αυτό ε, που γίνεται σε τοπικό επίπεδο θα πρέπει να διαφυλαχθεί, γιατί είναι θεμελιώδης δικαίωμα η πρόσβαση στο νερό. Θα πρέπει τη διαρμοδιότητα να βρίσκεται στους Δήμους και τις κοινότητες. Και αν ξεκινήσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης, ο εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα αυτό ήταν σαφής ότι θα πρέπει να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις αυτές. Και θα ήθελα να κάνουμε κάτι ενδιαφέρον εδώ. 20 ευρώ. 20 ευρώ σας δίνω αν μου πείτε, μια, αν μου αναφέρετε μια πολυεθνική που ενεργοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι ούτε, γερμα, ούτε γαλλική ούτε ισπανική. Στίχημα, άμα θέλετε. Γιατί όταν λέμε ότι, θα, θέλετε να απελευθερωθούν οι υδροδοτικέ εταιρείε, οι υπηρεσίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιο θα αποφεληθεί από αυτό. Σα δίνω 20 ευρώ αν μου αναφέρετε έστω και μια πολυεθνική που δεν είναι γαλλική ή ισπανική και ασχολείται με υπηρεσίε υδροδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στον επόμενο γύρο με εκπροσώπους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Αναφορών. Η Σοφία Κονίνη πρώτη στον κατάλογο. Για 1,5 λεπτό. Euh, Κυρίες και κύριοι, να χαιρετήσω κατά πρώτον την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών και την ακρόαση που σήμερα διοργανώθηκε, διότι επιτρέπει το θέμα του νερού να το θέσουμε στην καρδιά των ανησυχιών μας και ε, αυτό είναι πολύ θετικό. Ήδη εδώ και καιρό ε, αγωνίζομαι για τις πολιτικές χρηματοδοτήσεις και για την πρόσβαση όλων στο νερό και τα προκριτικά δίκτυα. τα σημεία 1 και 3 με βρίσκουν απολύτως σύμφωνοι μεταξύ όλων των υπολείπων που ούτως ή άλλως βλέπω θετικά ε, στη σημερινή μας συζήτηση για σήμερα το απόγευμα. Όμως για την απελευθέρωση των υπηρεσιών του νερού και όλες τις παρόμοιες κινήσεις που ανακοινώνονται σε σχέση με αυτό το θέμα. Οι υπηρεσίες καθαρισμού του νερού είναι στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από τις δημόσιες αρχές. Ένα τρίτο των Ευρωπαίων πολιτών επωφελούνται από αυτές τις ε, ε, υπηρεσίες ε, παροχής και καθαρισμού μέσω ιδιωτικών φορέων. Όμως να επιμείνω. Ακόμη και ένας δημόσιος φορέας είναι υπεύθυνο για αυτού του είδους την παροχή. Πάντοτε ε, ο ιδιωτικός φορέας θα βρίσκεται υπό την ε, παρακολούθηση του, του δημοσίου. Το να εκχωρηθεί λοιπόν ή να παραχωρηθεί μέρος της παροχής στα χέρια των ιδιωτών δεν είναι καθόλου αντίθετο με την προστασία αυτού του δικαιώματος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι άδικο να κατηγορούμε τις εταιρείες που έχουν αναλάβει δράσεις στον τομέα της ίδρευσης. Ενδιαφέρον θα ήταν σήμερα να ακούγαμε και το σύνολο των φορέων του χώρου που, της υδροδότησης συμπεριλαμβανομένων των εταιρεών υδροδότησης βασικές εταιρείες που εμπλέκονται στην, τομέα, στην ίδρυυση ε, είναι εταιρείες που συμβάλλουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία της. Επίσης, ε, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους επιτρέπει τη μείωση του κόστους και των τιμών επιτρέποντας να διασφαλίζεται και ποιότητα χωρίς αυτό να το χάνουν από τα χέρια του οι δημόσιες αρχές. Συμμετέχουν στην δημιουργία ΑΕΠ της χώρας μας, στην κερδοφορία και στην ανταγωνιστικότητά μας στις παγκόσμιες αγορέ. Μόνο οι ιδιωτικέ εταιρείε μπορούν μαζικά να επενδύσουν στην, στην καινοτομία και την έρευνα στον τομέα του νερού και βεβαίω αυτό είναι προφανέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. ευχαριστώ κυρία Κονή. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποιο συναδέλφους να διευκρινίσουμε δίτρα από την Επιτροπή ΙΜΚΟ ότι θα πρέπει να τηρούν το χρόνο της ομιλίας του. Σας παρακαλώ να τηρήσουμε το χρόνο ομιλίας γιατί δάλλως θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ο κ. Κρετονασένης, 1,5 λεπτό. Thank you, President. Ευχαριστώ. Η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι επιβλαβής ε, ε, κοινωνικά, παράλογη οικονομικά και δεν ε, στέκει και νομικά και ξεκίνησε από την πρωτοβουλία της κυρίας Θάτσερ που ιδιωτικοποίησε εταιρείε υδροδότησης και κάτι που οδήγησε σε αύξηση του, της τιμής του νερού για τους πολίτες. Είχαμε τριπλάσιο ρυθμό πολιτών που δεν είχαν πρόσβαση στο νερό γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ε, το, της ε, εταιρείας του νερού. Και στη Βολιβία η ιδιωτικοποίηση του νερού ε, οδήγησε της εταιρείε θα θέλουν να φορολογήσουν και τη συγκέντρωση των βρόχινων υδάτων. Πάνω από 2 εκατομμύρια, ε, λέμε, ε, Ευρωπαίων πολιτών πιστοποιημένα που έχουν υπογράψει κατά της ιδιωτικοποίησης της ίδρυυσης και μάλιστα και οι ευρωβουλευτές έγραψαν επιστολή ζητώντας από πολυεθνικές να καταλήψουν την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΔΑΠ Θεσσαλονίκης και μάλιστα ε, το Συμβουλίο της Επικράτειας ε, ε, ακύρωσε τη διαδικασία ιδιωτικοποίηση κρίνοντας την παράνομη. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί αυτή την παράλογη και παράνομη ιδιωτικοποίηση υπό το πρόσχημα των μεταρρυθμίσεων και υπό την αιγίδα και την ευλογία των εκπροσώπων της Τρόικα, στην οποία συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Σεύτσοβιτς. Έχουμε 15 εκατομμύρια αποθεματικό στην ΕΔΑΠ Θεσσαλονίκη, 18 εκατομμύρια κέρδη, πολλά εκατομμύρια ευρωπαϊκών επενδύσεων και το τίμημά της είναι 110 εκατομμύρια ευρώ. Και μάλιστα οι πολυεθνικέ το θεωρούν και υπερβολικό αυτό το τίμημα. Ζητώ από την ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει αυτή την παράνομη ενέργεια και ζητώ από τον Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Σευκοβίτση, να μου πει αν θέλουμε να σεβαστούμε του Ευρωπαίου πολίτε που μαζικά έβαλαν την υπογραφή του σε αυτή την πρωτοβουλία, θα πρέπει όταν επιστρέψετε στο γραφείο σα να πάρετε το τηλέφωνο και να ζητήσετε με του εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής στην Τρόικα και να του ενημερώσετε τέτοιε πολιτικέ δεν είναι πια ευπρόσδεκτε. Ευχαριστούμε, Κορίν Λεπάζ, για 1,5 λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που συμμετέχω σε αυτήν την ε, ακρόαση. Είναι ανδιαφυσβήτητη πρόοδος και είναι η πρώτη μέρα, το νούμερο ένα της δημοκρατίας των πολιτών στην Ευρώπη. Ελπίζουμε να υπάρχουν και άλλες τέτοιες πολλές ημέρες. Το να ακούει κανείς είναι καλό, αλλά το να παρακολουθεί αυτό που ακούει είναι ακόμη καλύτερο. Πρέπει λοιπόν η πρωτοβουλία των πολιτών, όπως διοργανώθηκε σήμερα, να εισακουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει οι κοινέ απόψεις που ακούστηκαν από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου και αυτές που εκφράστηκαν στην πρωτοβουλία των ε, πολιτών είτε μέσω της ε, πρότασης για τις παραχωρήσεις και του ψηφίσματός μας το 2012 όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Όμως υπάρχει αντίσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτές τις απόψεις και υπάρχει βούληση να προχωρήσει στο δρόμο της απελευθέρωσης. Απελευθέρωση την οποία δεν επιθυμούν πάρα πολλοί από του πολιτέ μα. Ναι, ίσως έναν ιδεατό κόσμο κόσμο να υπήρχε πραγματικό σωστό έλεγχο, να υπήρχε ισορροπία μεταξύ των ιδιωτικών εταιριών και του δημόσιου φορέα. Αλλά δεν βρισκόμαστε σε κόσμο ιδανικό και δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Εάν δει κανεί την αύξηση των τιμών του νερού, εάν σκεφτεί ότι το δημόσιο σύστημα και το ιδιωτικό ε, μπορεί να συγκριθούν μεταξύ του, θα το δούμε με πολλά παραδείγματα σε πολλέ χώρε, θα πρέπει να ακούσουμε του ε, περισσότερου από του Ευρωπαίου πολίτε που μα λένε ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν σε αυτή την Και δεν θα υπάρξει πραγματική ισορροπία. Ε, κυρία Πρόεδρε, Κυρία κύρια και κύριοι, δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ε, ε, συνέχιση της ε, απελευθέρωσης. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών. Σας ευχαριστώ, Μάρτιν Κέσλερ. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν ε, που δραστηριοποιηθήκατε. Θα ήθελα να σας συγχαρώ που συλλέξετε τόσες πολλές ε, ε, υπογραφές και καταδείξατε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη Γερμανία. Ακόμα και αν μεγάλος αριθμό των υπογραφών ήταν από τη Γερμανία, να σας πω ότι εμείς στη Βαυαρία έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες σε δημοτικό επίπεδο διοργανώνονται πάρα πολύ καλά και παρέχουν καθαρό νερό. Δεν χρειαζόμαστε ουσιαστικά ανταγωνισμό, χρειαζόμαστε ασφάλεια για τον πολίτη για να υπάρχει υψηλής ποιότητας καθαρό νερό. Αυτό είναι το καθαριστικό και γι' αυτό λοιπόν σας υποστηρίζω απόλυτα. Όταν μιλάτε λοιπόν για ε, διαφάνεια και για ανταγωνισμό, πάντα υπάρχει ένα επιχείρημα όσοι έχουν ευκαιρίες στην ιστορική αγορά και βλέπουμε λοιπόν στη σημερινή συζήτηση ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι όμιλοι με διάφορα συμφέροντα. Φυσικά λοιπόν αυτοί οι όμιλοι θέλουν να διευρυνθεί η αγορά. Αλλά οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι, οι πολιτικοί, οι δήμαρχοι, τα δημοτικά συμβούλια που δραστηριοποιούνται για να υπάρχει σωστή παροχή νερού, αυτοί θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Αυτοί θα πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις και θα πρέπει λοιπόν ο τομέας της αγοράς να συνεχίσει να εξαιρείται και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το TTIP, τη συζήτηση για την ζωνή ελευθερού με την Αμερική. Λοιπόν, τι να σας πω, στην υγειά σας. uns heute. Μάλιστα λοιπόν, ε, υψώνει το ποτήρι ο συνάδελφος από τη Βαβαρία. 1,5 λεπτό η επόμενη μιλήτρια. Κυρία Νέσα Τσάιλντερς, ευχαριστώ. Αυτή η εκστρατεία για το δικαίωμα στο νερό είναι πολύ επίκαιρη. Πολλά δε μάλλον που πολλέ χώρε όπω η πατρίδα μου η Ιρλανδία εφάρμοσαν τέλη νερού και έχουν, και, και έχουν ε, ε, στα πλαίσια του πακέτου διάσωση έχουν ιδιωτικοποιήσει ένα τμήμα του τομέα. Και μάλιστα στο μέλλον θα έχουμε υψηλότερου λογαριασμού νερού και χειρότερε Υπηρεσίε και κακής ποιότητας. Οι πολίτες μας που έχουν πληγεί από, και από την κρίση και από τις πολιτικές λιτότητας ε, θα δεν θα μπορούν πια να πληρώνουν αυτά τα δικαιολόγητα ψηλά και ανήθικα τέλη για το νερό εξαιτία τη ιδιωτικοποίηση. Θα πρέπει να προσέξουμε όλα τα στάδια από την παραγωγή στην κατανάλωση και να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα είδωρ. Επίση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τον έλεγχο στην πρόσβαση στο νερό, που είναι δικαίωμα για όλου του πολίτε. Δεν θα πρέπει να ε, απελευθερώσουμε την πρόσβαση στο νερό και να το καταστήσουμε εμπορικό προϊόν θα πρέπει να είναι προσιτές οι τιμές του νερού και να είναι προσιτό σε όλους και να είναι και ποιοτικό. Μόνο όταν όλοι έχουν δικαίωμα και πρόσβαση στο νερό θα έχει πραγματικά το καθεστώς ανθρώπινου δικαιώματος. Το θέμα των τιμών, πώς θα εξασφαλίσετε ότι θα υλοποιήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και την οικουμενική πρόσβαση στην ίδρυυση και στην αποχέτευση. Επίσης, τι μέτρα θα θεσπίσετε ώστε να βελτιώσετε τη συμμετοχή των χρηστών και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία διαδικασία λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο νερό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χουντής. 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, είμαι Ευρωβουλευτής από την Επιτροπή Αναφορών, από την Αριστερά και από την Ελλάδα. Συγχαίρω την προσπάθεια που γίνεται. Η προσπάθεια και αυτή η πρωτοβουλία είναι αξιέπαινη, όμως με αφορμή και το παράδειγμα της Ελλάδας που ήδη αναφέρθηκε αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται και με άλλες μορφές, καθώς γνωρίζετε ότι η απόπειρα ιδιωτικοποίησης των δικτύων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη συναντά τις μαζικές αντιδράσεις των πολιτών, ζητούν να αποφασίσουν με δημοψήφισμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα, αναφέρθηκε. Η, Επιτροπή, η Κομισιόν δείχνει ευαισθησία. Απάντηση του κυρίου Μπαρνιέ. Το νερό έξω από την οδηγία παραχώρησης. Απάντηση του κυρίου Ρεν το νερό και η ιδιοκτησία στα δίκτυα δεν το πιέζουμε εμείς να αλλάξει και να μην είναι δημόσιο. Αποτέλεσμα όμως, μέσω της Τρόικα η ελληνική κυβέρνηση τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται ότι τις επιβάλλουν και προχωράει στο ξεπούλημα των δικτύων ίδρυυσης και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ερώτηση, επειδή γίνεται ένας διάλογος, ερώτηση τον κύριο Ρεν. Μπορείτε να μου πείτε το βίο και την πολιτεία το βίο και την πολιτεία των μεγάλων πολυεθνικών μονοπωλίων της ίδρευσης που εμφανίζονται ως αναλλακτικέ λύσεις για να εξαγοράσουν τα δίκτυα. Καμία απάντηση. Επομένως, ο αγώνας για να υπερασπιστούμε το νερό ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα πρέπει να συνοδεύεται από την προσπάθεια να κατοχυρωθεί ως δημόσιο αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye και έχω δύο μιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο, η Evelyn Γκέπχαρτ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Μιλώ τώρα εξ ονόματος του συναδέλφου Αντώνιου Πανθενή, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί και μου ζήτησε να θέσω μια ερώτηση εξ ονόματος του από την οδηγία για τη συμβάση παραχώρησης που είναι και εισηγητής ο συναδελφός μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταφέραμε να βγάλουμε τον τομέα του ύδατος. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ικανοποιείται, δεν είναι καθόλου ευχαριστημένη με αυτό και αυτό είναι γεγονός. Ερωτώ λοιπόν, τι θα γίνει τώρα, πώς θα συνεχιστεί η κατάσταση. Πώ θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει. Κάποιοι είπαν ότι ναι, σε δύο-τρία χρόνια θα εξετάσουμε πώ θα έχει η κατάσταση. Όντω, θα ξεκινήσετε από την αρχή αυτή τη διαδικασία ή μήπω σε κάποια στιγμή μπορεί να μπει μία τελεία και να πούμε ότι είναι ένα κοινό αγαθό το νερό. Δεν είναι εμπόρευμα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εμπορευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εύελεν Κέπχαρτ, λέει ο πρόεδρο, Ένα λεπτό ακριβώ Και η κυρία Κουτιέρε. Ευχαριστώ. Φοβάμαι ότι δεν είναι ακριβείς όλες οι πληροφορίες που ακούσαμε. Γιατί άλλο να είναι το νερό δημόσιο αγαθό και τα δίκτυα να είναι δημόσια και άλλο θέμα είναι η ιδιωτική διαχείριση. Είπαμε ότι θέλουμε διαφάνεια. Έχουμε πολλούς δήμους που σε συμφωνία με ιδιωτικούς φορείς οι ίδιοι οι δήμοι καρπώνονται ένα μεγάλο τμήμα των εσόδων από το νερό και μάλιστα το χρησιμοποιούν ως μαύρα κονδύλια των δήμων. Ξέρω ευρωπαϊκούς δήμους που εισπράττουν 300 και 400 εκατομμύρια ε, ευρώ από τις εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει τις παραχωρήσεις και μετά διαχειρίζονται αυτά τα κονδύλια ως μαύρα κονδύλια του προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλούμε για δημόσια διαχείριση αν δεν έχουμε σωστή νομοθεσία που θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια, κάτι που δεν έχουμε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γιατί ε, δεν ξέρουμε από πού έρχεται το νερό, ε, γιατί είχαμε αντίστοιχο παράδειγμα και με τον ηλεκτρισμό. Θέλουμε λοιπόν καλή πρωτοβουλία, αλλά να ρυθμίσουμε το θέμα της διαφάνειας, της ετοιμότητας και να μην ε, παραπλανούμε τους πολίτες λέγοντας απλώς ότι είναι δημόσιο αγαθό. Γιατί μερικές φορές ε, γίνεται κακή διαχείριση και από το δημόσιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα περνάμε στην απάντηση των ερωτήσεων που ακούσαμε από την Επιτροπή των Πολιτών. Οκτώ λεπτά για τη διάθεσή σας και επιλέξτε εσείς ποιος θέλετε να μιλήσει. Ο κ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι εγώ δεν θα χρειαστώ και πάρα πολύ χρόνο. Δύο στοιχεία θα ήθελα στο να τονίσω γιατί είναι ζωτική σημασία. Το θέμα της διαφάνειας και το θέμα αυτό το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ κέριο είναι από πού προέρχονται τα κέρδη, πόσο υψηλά είναι τα κέρδη, ποιον ωφελούν. Του ιδιωτικούς μετόχους, των δημοσίων εταιριών υδροδότηση, ποια είναι η επενδυτική σχέση σε ό,τι αφορά τη δημιουργία, την, ε, τον εξυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Εδώ θεωρώ ότι λείπουν πολλά και θα θέλαμε η οδηγία για τη διαφάνεια να προδιαγράψει το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται και οι ιδιωτικοί φορείς. Ότι θα πρέπει να υπάρχει κέρδος είναι κάτι το μη αμφιλεγόμενο. Στην πόλη στην οποία ζω το έχουμε δει. Με δύο, με την ε, εταιρεία υδροδότησης ε, του Βαρολίνου, με τη συμμετοχή δύο ιδιωτικών μετόχων η πόλη, ο Δήμος εκχώρησε τα δικαιώματά του για κέρδος υπέρ των ε, ιδιωτικών μετόχων που έπρεπε να έχουν κάποιο εγγυημένο ποσοστό κερδών. Αυτό δεν επιτρέπεται λοιπόν να συνεχιστεί. Και αυτό είχε και συνέπειες σε ό,τι αφορά παροπλισμό παλιών εγκαταστάσεων, σε ό,τι αφορά ε, τις συνέπειες, τις περιβαλλοντικές για τον υδροφόρο ορίζοντα. Γιατί κοιτάξτε το θέμα της ε, υδροδότησης δεν είναι μόνο θέμα υδροδότησης, έχει να κάνει και με άλλα ζητήματα πέρα από την αμυγή υδροδότηση σε ό,τι αφορά το θέμα της απελευθέρωσης και τον ανταγωνισμό όταν συμμετέχει και μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ανταυτό τι γίνεται. Η υδροδότηση λέμε ότι αποτελεί φυσικό μονοπόλιο. Και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ε, ιδιωτικός Αν οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αναγκαστούν να, κάνουν, να βγάλουν κέρδη, θα μπορέσουν μέσω των τελών για την εθοδότηση να συλλέξουν τα μέσα προκειμένου να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις. Υπάρχει λοιπόν ένας, μια βασική διαφορά την οποία θα πρέπει να τη λάβουμε υπόψη. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό από αυτά που έως τώρα έχουμε ακούσει. Ε, Tommaso Fattori, Forum Italiano Movimento. Ε, λέγομαι το Μάζο Φατόρη και εργάζομαι. Τα πολλά να πω ότι για την πρωτοβουλία των πολιτών δεν υπάρχει καμία σύγχυση μεταξύ των υπηρεσιών και του ίδιου του νερού φυσικού πόρου. Ε, πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε το φυσικό αγαθό, το νερό ε, και τις υπηρεσίε παροχής του εάν θέλουμε να το εγγυηθούμε το δικαίωμα της πρόσβασης στο νερό ως ένα θεμελιώδης δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και τα δύο λοιπόν στοιχεία είναι αλληλένδετα, δεν μπορούν να διαχωριστούν ε, και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό και η πρόσβαση σε αποχετευτικά δίκτυα. Τώρα, για τα καθοριστικά στοιχεία της πρωτοβουλίας μας, δεν μπορούν να διαστρεβλώνονται με το επιχείρημα της επικουρικότητας ή με πρόσχημα αυτό το επιχείρημα. Πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να πάυσει αμέσως η σημερινή τάση προς την απελευθέρωση. Μία τάση και μια όθηση που έρχεται πραγματικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι επίσημη συνιστόσα τη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το έχουμε ήδη πει. Εάν δούμε τι ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Πορτογαλία, αυτή είναι η υποχρέωση. Πρέπει να απελευθερώσετε τι υπηρεσίε ίδρυψή σα, εάν θέλετε την ενίσχυση από τα ταμεία διάσωση, ε, από τα κονδύλια τα δικά μα. Δηλαδή, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρησιμοποιεί αυτό τότε επιχείρημα για να δώσει χρήμα στις χώρες του Νότου και τώρα το χρησιμοποιεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν, εάν δεν αναγνωρίσουμε ρητός το ε, δικαίωμα πρόσβαση στο πόσιμο νερό και στις αποκαιτευτικέ υπηρεσίες ως ένα νομοθετικό δικαίωμα, ένα δικαίωμα νομοθετημένο, θεσμοθετημένο μέσα από την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον αυτό δεν γραφεί επί χάρτου, δεν θα υπάρξει προστασία του νερού. Κανένα πολίτη δεν πρέπει να αποκλείεται από την πρόσβαση στο νερό. Ανάληψη τη ευθύνη σημαίνει ότι θα βρούμε και ειδικά κονδύλια για επενδύσει που επιτρέπουν την πρόσβαση όλων, την οικουμενική πρόσβαση στο νερό. Ακόμα και από τι φτωχότερε περιοχέ τη Ευρώπη που δεν είναι εύκολο αυτό. Υπάρχουν όλο ένα και περισσότερε οικογένειε των οποίων το εισόδημα μειώνεται λόγω τη κρίση και μπορεί να βρεθούν εκτό παροχή υπηρεσιών. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί η φτώχεια να είναι λόγο για να αποκλείεται αποκλείεται κανείς από το δικαίωμα ίδρυυσης. Δεν μιλάμε για αγορά, δεν μιλάμε για χρήμα και εμπόριο, αλλά για ζωή. Εδώ λοιπόν απαιτούμε ένα πλαίσιο. Κάτι που έρχεται και πριν καν από τη συζήτηση για την απελευθέρωση και την ιδιωτικοποίηση. Προτεραιότητα για τι ευρωπαϊκέ πολιτικέ του νερού θα πρέπει να είναι η προστασία τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη ανθρώπινη ζωή, όχι η υγεία των αγορών και των εμπορευομένων. Ξέρουμε ότι δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το αν η ίδρευση και η παροχή νερού θα είναι δημόσιο ιδιωτικό ζήτημα στα επιμέρους κράτη-μέλη, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά ζητούμε ένα πλαίσιο, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και τουλάχιστον να αποκλειστεί υποχρέωση απελευθέρωσης. Μιλάμε για ένα στοιχείο δημοκρατίας. Οπουδήποτε εκφράστηκαν για το θέμα αυτό οι πληθυσμοί, οι πολίτε τη Ευρώπη τάχθηκαν κατά τη ιδιωτικοποίηση. διότι τα αποτελέσματα τη ιδιωτικοποίηση, στις περισσότερε χώρε ήταν καταστροφικά. Έγιναν τρία δημοψηφίσματα σε τρει χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τρεις πόλεις Ευρωπαϊκή ε, Ένωση στην Ιταλία και αλλού και κάθε φορά οι πολίτε τάχθηκαν κατά, κατά και των ιδιωτικοποιήσεων. Αλλά α πούμε ότι τουλάχιστον γνωρίζουμε το δικαίωμα στο νερό και ότι λέμε όχι στι διαδικασίε απελευθέρωση που έρχονται από πάνω από αλλού και αν δώσετε το δικαίωμα στους πολίτες να αποφανθούν θα δείτε ότι σας πούνε ένα ηχηρό όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Πολύ σύντομα θα ήθελα να απαντήσω στη Γαλλίδα Ευρωβουλευτή φαίνεται ότι υποστηρίζετε τις ιδιωτικές ε, εταιρείε ίδρυυση, ε, γιατί τα ίδια επιχειρήματα θα μπορούσαν να ισχύουν και για τι ε, δημόσιε. Εμεί δεν είμαστε για τι ιδιωτικέ, δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Απλώ ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην απελευθερώσει τι υπηρεσίε ίδρυυση. Ενώ το δικό σα κόμμα είναι υπέρ τη απελευθέρωση των αγορών και στον τομέα του ύδατο. Οπότε ζητούμε δέσμευση νομοθετική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην απελευθερώσει τις, ευρωπαϊκές, τις υπηρεσίες ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον κύριο Τζόναθαν Φόλ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης ε, Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ αγαπητοί Ευρωβουλευτές. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτη και ιστορική αυτή η στιγμή και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την οργάνωση. Κάποιες παρατηρήσει για να διασκεδάσω κάποιες αφιβολίες και να διορθώσω για κάποιες παρεξηγήσεις. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες για τις παραχωρήσεις η Ευρωπαϊκή, Υπηρεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι, όχι μόνο δεν ήταν δυσαρεστημένη, αλλά ήταν και υπερβολικά ικανοποιημένη με την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Και έχω και τη δήλωση της 21ης Ιουνίου του κυρίου Μπαρνιέ, που λέει ότι η καλύτερη λύση φαίνεται ότι είναι να αφαιρεθεί το νερό από το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία για τι παραχωρήσει. Θα πρέπει, για καθήκον μα, να λάβουμε υπόψη τι ανησυχίε ε, πολυάριθμων συμπολιτών μα. Και θα προτείνω στον πρόεδρο Μπαρόζο και στου υπόλοιπου επιτρόπου να επικυρώσουν αυτή τη διαδικασία, την απόφαση, όπω και έγινε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυ, την κατάσταση στον τομέα ύδατο. Αυτό. Αυτά ως τώρα, τα θέματα τη αναθεώρησης και τις σχετικέ ανησυχίες που εκφράστηκαν, είναι σαν ε, είναι ένα σήμα ότι από κάποια κερκόπορτα θα ανακληθούν αυτές οι αποφάσεις, σας διαβεβαιώ ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά θα πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει στα κράτη-μέλη. Πάντως είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η, η θεμελιώδης δημοκρατική απόφαση για την οργάνωση της παροχής ύδατος είναι μια απόφαση που λαμβάνεται τοπικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία αρμοδιότητα και καμία εξουσία να ε, επιτάξει, να υποδείξει ότι το είδωρ θα πρέπει να παρέχεται με, από δημόσιους ιδιωτικούς φορείς και ούτω καθεξής. Γιατί αυτό φαίνεται να ακούσαμε από διάφορους. Αυτά είναι αρμοδιότητες και εξουσίες δημοκρατικών και τοπικών επιλογών που γίνονται, που αναθεωρούνται, αλλάζουν. Πάντως ε, Ίσως σε μία πενταετία θα έχουμε νέα αναθεώρηση, κάτι που γίνεται σε περίπλοκες ε, νομοθετικές πράξεις. Θα επανεξετάσουμε την κατάσταση και θα ενημερώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ενημερώσουμε και το Συμβούλιο και θα λάβουμε φυσικά υπόψη και την συνέχεια που θα δοθεί, που σίγουρα θα υπάρξει μετά από πολύ σημαντική ιστορική σημασίας πρωτοβουλία της ε, πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν μπορώ να προβλέψω τώρα τι θα πει, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από μία πενταετία. Πάντως ε, μπορώ βάσιμα να προβλέψω ότι θα λάβει σίγουρα υπόψη το κίνημα που δημιουργήθηκε με την πρωτοβουλία αυτή και θα λάβει υπόψη και την συνέχεια της συζήτησης που θα διεξαχθεί στα κράτη-μέλη. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει η οδηγία για τις παραχωρήσεις και θα ενημερώσουμε σχετικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τώρα, για άλλα θέματα και επανέρχομαι στο γενικό θέμα της απελευθέρωσης του τομέα ύδατος. Μπορεί να δηλώσει κατηγορηματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει κανένα σχέδιο να απελευθερώσει την ίδρυυση, την παροχή ύδατος. Καταρχήν εξαρτάται από τον ορισμό που θα δώσουμε στην απελευθέρωση και συμφωνώ με όσους είπαν ότι η απελευθέρωση δεν είναι συνώνυμο της ιδιωτικοποίησης. Και κυρίως αυτό το θέμα επαφίεται στα κράτη-μέλη. Αν ένα κρατος μέλος ή ε, μια περιφέρεια με βάση τις, ε, τους δημοκρατικούς και συνταγματικούς κανόνες ε, κρίνουν ότι το, νερό θα πρέπει να παρέχεται με τον ΑΒ τρόπο, το κράτος μέλος είναι κυρίαρχο να κάνει κάτι τέτοιο. Αν μια χώρα αποφασίσει να κρατήσει το νερό, τη διαχείριση και την παροχή ύδατος στα χέρια του δημοσίου και να απομονώσει αυτά τα θέματα από την αγορά και πάλι έχει τη διακριτική ευχαίρεια να το κάνει το κράτος μέλος και πολλές χώρες ε, το έχουν κάνει. Ούτε στο θέμα αυτό έχουμε κάποιο λόγο. Και η συνθήκη μας υποχρεώνει να μην έχουμε λόγο στα θέματα αυτά. Τώρα, άλλη απόφαση, όπως είναι σε άλλες χώρες, μετά από συζήτηση φυσικά και επανεξέταση αποφασιστεί να ανοίξουν κάποια στοιχεία της παροχής ύδατος ε, στους κανόνες της αγοράς, να γίνει μια απελευθέρωση, όπως έχει συμβεί. Και αυτό ε, γίνεται, γιατί η εσωτερική αγορά καλύπτει όλα τα κρατημέλη, οπότε σε τέτοια περίπτωση ισχύουν οι κανόνες της διαφάνειας, η αποφυγή των διακρίσεων και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό είναι ε, ε, αυτό που πυροδοτεί η, την απόφαση. Είναι θέμα τοπικής εθνικής απόφασης και όχι ευρωπαϊκής απόφασης. Η δημοκρατία λαμβάνει χώρα και σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. Εμείς απλώς σημειώνουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο κατάλληλο επίπεδο. Επαναλαμβάνω τη δήλωση και τις δράσεις του Επιτρόπου Μπαρνιέ και την ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για να αποφευθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, αφαιρούμε το είδωρ από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας για τις παραχωρήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανένα απολύτως σχέδιο να κάνει περαιτέρω ενέργειες ε, προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης, όπως λέτε, σε ό,τι αφορά την παροχή του ύδατος. Εμείς θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σε όλα τα κράτη-μέλη και θα αντιδράσουμε αν το αργότερο σε μία πενταετία τότε που θα γίνει και η αναθεώρηση της οδηγίας για τις παραχωρήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κλείνοντας ο κύριος Ότου. Σας ευχαριστώ πολύ. Είπατε πριν από λίγο ότι δεν ξέρετε πώς, ε, πώς θα σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πέντε χρόνια. Ούτε εμείς το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν τώρα χρειάζεται να γίνει το βήμα. Να πούμε ότι αναγνωρίζουμε η υδροδότηση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και για, σε μόνιμο επίπεδο δεν πρόκειται να υπόκειται στις ε, ε, κανόνες της ε, αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν η συζήτηση η οποία γίνεται και ξαναγίνεται για το θέμα του ανοίγματο της αγοράς σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και την αποχέτευση είναι ακριβώς το πρόβλημα το οποίο επανεμφανίζεται επί 20 χρόνια, κάθε τρεις και λίγο. Και γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι τώρα θα πρέπει να γίνει το μη. Και νομίζω ότι αυτό θα το συζητήσουμε πάρα πολύ στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα με τους υποψήφιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστούμε κύριε Ότ. Και τώρα να περάσουμε στις καταληκτικές ε, δηλώσεις, παρεμβάσεις. Να καλωσορίσω δύο εκπροσώπους και από άλλα θεσμικά όργανα, τα οποία δεν έχουμε πάντα εδώ μαζί μας, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Η κυρία Νουάι Μαριέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ε, υποστηρίζουμε και είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και στηρίζουμε την πρωτοβουλία ώστε η πρόσβαση στην ίδρυυση και την αποχέτευση να καθιερωθούν ως ανθρώπινο δικαίωμα, όπως προβλέπει τα ε, από το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών και μετά το 2015 και να προβλέψουν παροχή ύδατος και αποχέτευσης ως ε, θεμελιώδη ε, κοινοφελής υπηρεσίες. Ανταποκριθήκαμε στην πρωτοβουλία της Ουγγρικής Προεδρίας για τη συμπερίληψη της πολιτικής του ύδατος στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πολιτικές και μάλιστα και σε μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εταιρική σχέση για την καινοτομία στο νερό και σε ένα σχέδιο δράσης για την διαφύλαξη των υδάτων πόρων στην Ευρώπη εκδώσαμε και και δημοσι... Ε, και μάλιστα είχαμε και την κυρία Καρόλα Μπαρς ε, ε, που είναι Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κοινοφελών Υπηρεσιών και την κυρία Χαλ Φέριχ, που είναι πρόεδρος της, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταπολέμησης της Φτώχειας στην, στην Ολομέλειά μας του Δεκεμβρίου γιατί εμείς υποστηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι για να θεσπίσουμε μια τέτοια νομοθεσία που θα καθιστά οικουμενική την πρόσβαση στο είδωρ και την αποχέτευση. Θα πρέπει να κάνουμε διάκριση μεταξύ των ε, και επικερδών υπηρεσιών, επιχειρήσεων που αποκομίζουν κέρδος από την υδροδότηση και από τη, ε, μεταξύ αυτών και των κοινοφελών υπηρεσιών που θέτει το είδωρ στην υπηρεσία του πολίτη. Επίσης θα πρέπει με διαφανή τρόπο να δούμε τα αποτελέσματα των μελετών που έγιναν από την ε, εταιρική σχέση για την καινοτομία για το είδωρ και να έχουν πρόσβαση σε αυτά και τοπικοί φορείς ε, και ε, άλλοι τοπικοί και οικονομικοί παράγοντες. Επίσης θέλουμε πόσιμο είδωρ που θα τη χάνει εύκολη επεξεργασία, γιατί δεν έχουμε πια φυσικό είδωρ. Επίσης θα πρέπει ο κατάλογος με τις υπογόνες ουσίες να διευρυνθεί, ώστε να ε, ξαναδούμε ποιο είναι το κόστος της ρήπασης και το κόστος της επεξεργασίας των υδάτων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην πολιτική γειτονία αλλά και στην εμπορική της πολιτική να λαμβάνει υπόψη την επίπτωση που έχουν τα μέτρα που λαμβάνει στην εξωτερική της πολιτική. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ και τώρα από την ε, Επιτροπή των Περιφερειών το λόγο έχει η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχά, χαρητήρια για του διοργανωτέ αυτή τη πρώτη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών και σα ευχαριστώ Πρόεδρε που, εφαρμο... που προσκαλέσατε την Επιτροπή των Περιφερειών σε αυτή τη συνάντηση. Πράγματι, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τι 7 πρώτε πρωτοβουλίε ε, των ε, πολιτών στην Επιτροπή των Περιφερειών με τον ε, πρόεδρο της Επιτροπής των Πρωτοβουλειών αυτών, τον κύριο Γκουντριάν. Και πρέπει να πω κατά πρώτον ότι οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να εμπλεχθούν στην διαχείριση, τη βιώσιμη διαχείριση της ε, και των υπηρεσιών ίδρυψης καθώ και των συμβάσεων παραχώρησης. Ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο τη θέση μας. Πρώτα απ' όλα το νερό είναι ένα αναπαροτρίωτο δικαίωμα, ένα δικαίωμα στη ζωή και ότι οι αρχέ ε, τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκησης μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο στον ε, διαχείρισή του. Το είπε και ο κύριος Κόλ από λίγο. Και επίσης χρειάζεται μια πιο υπεύθυνη συμμετοχή των ε, αρχών που είναι υπεύθυνε για την ίδρυυση στην διανομή του νερού, την παροχή του νερού και την ε, διαχείριση των αστικών λιμάτων. Θα πρέπει οι αρχέ αυτέ να ε, συμμετέχουν ενεργά στο μέλλον στην κατάρτιση τη μελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική για το νερό. Κατά δεύτερον, ε, είμαστε κατά της, του να υπόκειται το νερό στην αγορά, στην λογική τη αγορά δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό, θα πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση της ανθρωπότητας, καθότι είναι απαραίτητο για την επιβίωση των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων. Θα πρέπει λοιπόν οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση του νερού και ε, να αποκλειστούν από την οδηγία των συμβάσεων παραχώρησης και να καταρτιστεί σαφής πολιτική για την τιμολόγηση του νερού και των υπηρεσιών του. Θα πρέπει να αναλάβουμε το καθήκον μας, να σεβαστούμε το και να προστατεύσουμε από το φυσικό πόρο αυτό το ανεκτήμητο αγαθό για το καλό των πολιτών μας και των μελλοντικών γενναιών. Ευχαριστώ Πρόεδρε που προσκαλέσατε την Επιτροπή των Περιφερειών και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κουτριάν, ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Πολιτών, για να συνοψίσει και να προβεί και στα καταλητικά σχόλια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πολλοί το είπαν ότι συμμετέχετε, συμμετέχετε όλοι σας σε ένα ιστορικό γεγονός. Όντως είναι ιστορική αυτή η εκδήλωση, η πρώτη πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών που πέρασε το όριο και έθεσε ένα τέτοιο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Είναι ιστορική σημασία το γεγονός αυτό και για τη συμμετοχική δημοκρατία στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία για θέματα ε, περιβάλλοντος, φτώχειας, ε, ισότητας των γυναικών ε, τάσεται για όλα αυτά τα θέματα, αλλά και σε επίπεδο δημοτικό, όλος ο κόσμος έχει υποστηρίξει την ε, εκστρατεία μα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για την υποστηρίξή σας αυτή. Όσοι υποστήριξαν την πρωτοβουλία για το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό και στην αποχέτευση έχουν μια σαφή έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομοθετική πρόταση που θα εφαρμόζει τι υπηρεσίε όπω ορίζονται από το ψήφισμα του 2010 του ΟΗΕ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου ο κόσμος να έχει πρόσβαση αξιόπιστη σε υψηλής ποιότητας νερό και αυτό αποτελεί σημαντική προϋπόθεση και για την εξωτερική πολιτική αλλά και για την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί συνάδελφοι και πολλοί βουλευτές τόνισαν πόσο θετική είναι η επιρροή σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θέματα ύδατο και αποχέτευση σε όλο τον κόσμο. Επίσης, πολλοί από του υποστηρικτέ μα υποστηρίζουν την έκκληση η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να μην υπόκειται σε κανόνες της αγοράς και ότι δεν θέλουν αυτές οι υπηρεσίες να απελευθερωθούν. Υποθέτω ότι σε πέντε χρόνια όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μάλλον το να σκεφτόμαστε και να εικάζουμε το τι θα συμβαίνει σε πέντε χρόνια δεν αρκεί. Θέλουμε να μην υπάρξει απελευθέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υπηρεσιών αυτών και αυτό τονίζουμε, αυτό υπογραμμίζουμε ότι δεν θέλουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σαφές και ξεκάθαρο ως έκκληση και ως απέτηση. Το νερό λοιπόν δεν αποτελεί ένα εμπόρευμα, είναι ένα δημόσιο αγαθό, είναι η ζωή και αυτό το διακηρύσει και το ιστοσελίδα της ε, γενική διεύθυνση περιβάλλοντο, Είναι ένα πολύτιμο αγαθό το οποίο θα πρέπει να διαφυλάξουμε και για τις μελλοντικέ γενιές. Εμεί και η πρωτοβουλία μας θέλουμε να γνωριστεί το νερό και οι υπηρεσίε αποχέτευση ως κάτι θεμελιώδες για την ευημερία μας, για την οικονομία μας, για το περιβάλλον μας. Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Δικαίωμα στο Νερό έχει υποστηριχθεί από πολλά εκατομμύρια πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλοί από τα συνδικάτα, από, σύμφωνη από συνεδριάσεις ε, διάφορων οργανώσεων Πολλοί βγήκαν στους δρόμους, πήγαν σε εμπορικά κέντρα για να συλλέξουν ε, υπογραφές. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την υποστήριξη αυτή και η Επιτροπή α, των Πολιτών και όλοι εμείς σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη εξ ονόματος όλων των πολιτών που υπέγραψαν, που προσυπέγραψαν την ε, έκκληση. Τώρα ε, το θέμα είναι να ανταποκριθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει την ευκαιρία να καταδείξει το τι θεωρούμε ότι είναι η ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τοποθετηθεί στο επίκεντρο των δράσεών μας ο άνθρωπος. Να κάνουμε κάτι για τις μελλοντικέ γενιές. Έχει την ευκαιρία να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων των υπεύθυνων της πρωτοβουλίας, κάλλοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μας απογοητεύσει, να δράσει και να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει το αίτημά μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν την συνεδρίαση αυτή και πολλοί κόσμος αλλά και πολλοί βουλευτές ε, είπαν ότι έχουμε λόγο να γιορτάσουμε σήμερα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε και κάποιο λόγο να γιορτάσουμε σήμερα, αλλά όταν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκριθεί στο αίτημα των πολιτών, τότε θα έχουμε τον πραγματικό λόγο να γιορτάσουμε και τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία αποτελεί πραγματικά ένα εργαλείο συμμετοχικής δημοκρατίας και όχι κάτι το οποίο μπορούμε να ξεπετάξουμε και να παραγωνίσουμε αν το επιθυμούμε. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλούμε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δράσετε αναλόγως. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκούρντιαν για το καταληκτικό σας αυτό σχόλιο και θα ήθελα τώρα να δώσω τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το λόγο για να κάνει και αυτό τα καταλητικά του σχόλια. Σε ό,τι αφορά και το μέλλον, ελπίζουμε να γίνουν αυτά πριν από την Παγκόσμια ημέρα, ημέρα του νερού, 22 Μαρτίου. Έχετε το λόγο κύριε Σεφκοβίτσο. Ευχαριστώ πολύ Ματέας. Ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε τόσο πολύ ε, εδώ. Ευχαριστώ για την αθροά προσέλευση λοιπόν και ευχαριστώ και την Διοργανωτική Επιτροπή για αυτή την εξαιρετική ακρόαση. Είδαμε πόσοι πολλοί είστε εδώ, τι καλή γεωγραφική κάλυψη είχαμε και τι ενδιαφέροντα θέματα συζητήθηκαν στην ατζέντα. Παρόλο που ήταν μακρά η ημέρα αυτή και η συζήτηση κράτησε πολύ, νομίζω ότι με τη συζήτηση ακριβώς είδαμε ότι η πρωτοβουλία είναι, να ευρύτα το θέμα. Ένα θέμα που ε, το συζητήσαμε και το πρωί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα το συζητάμε στο Ευρωκοινοβούλιο, Όλους μας αφορά ιδιαίτερος. Προφανώς για μένα και τους συναδέλφους μου είναι πολύ σημαντική συνάντηση, διότι καταγράψαμε τις λεπτομέρειες των τοποθετήσεών σας για να δούμε τι συγκεκριμένες πτυχές πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο μας καλέσατε επανειλημμένως σε δράση και πραγματικά σας το λέω ότι θα το κάνουμε εν ευθέτω χρόνο διότι όπως και εσείς σεβαστήκατε όλους τους κανόνες και τους ε, που είχαμε ορίσει εμείς και τα κριτήρια το ίδιο θα κάνουμε και εμείς θα αναλύσουμε όλες τις πτυχές της πρωτοβουλίας και θα φροντίσουμε τα συμπεράσματα να σας τα υποβάλουμε σύντομα. Όχι σήμερα, γιατί θέλησαμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις, τις διακλαδώσεις τους και να σεβαστούμε και τους περιορισμούς που υπάρχουν λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά θα φροντίσουμε να ε, δημοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση το αργότερο στις 20 Μαρτίου. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ορισμένα σημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για μένα. Άκουσα την έκκλησή σας για περαιτέρω αναγνώριση του ε, νερού ως ανθρωπίνου δικαιώματος το θέμα είναι πώς να υλοποιηθεί ακριβώς η προστασία του δικαιώματος αυτού. Πώς να υπάρξει μια κοινή κατανόηση ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τις εκκλήσεις σας για το ότι πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο την αναπτυξιακή μας πολιτική προς αυτή την κατεύθυνση. Ακόμη και για τα προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και θα γνωρίζετε φαντάζομαι πόσα κάναμε ήδη σε αυτό το τομέα, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα και ακούω αυτά που λέτε. Επίσης για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την διαφανέστερη συμπεριφορά, την καταγραφή των επιδόσεων των εταιριών παροχή ύδατο ανά την Ευρώπη. Αυτό είναι σαφέ. Ενδιαφέρει όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλουν να ξέρουν πώ τα πάνε αυτέ οι εταιρείε, τι κέρδο έχουν, τι κάνουν το δημόσιο χρήμα και τι πληρώνουν ακριβώ οι πολίτε για τι υπηρεσίε που λαμβάνουν. Πώ ξοδεύετε το χρήμα τους. Ταυτόχρονα να σας πω ότι δεν είναι απλό ε, αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρωτοβουλία σας καλύπτει μια σειρά από πολύ διαφορετικά θέματα. Θα πρέπει διαφορετικές γενικές διευθύνσεις να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια. θα καλυφθούν όλα αυτά τα ζητήματα στην ανακοίνωση της 20ης Μαρτίου. Θα πρέπει λοιπόν με όλες τις γενικές διευθύνσεις να δούμε πώς θα προσεγγίσουμε την δική σας πρωτοβουλία και θα φροντίσουμε να το κάνουμε καλόπιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά ένα-δυο ένα, δυο ενα ζητήματα που εφήγησαν. Ε, για τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών. Νομίζω το συζητήσαμε και το πρωί. Όμως, θα το παραλάβω και εδώ. Εάν μιλάμε για τις κοινοφελείς υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντοτε είναι πολύ προσεκτική για το πώς αυτά συμπεριλαμβάνονται στη διαπραγματευτική της αντολή και πώς τα διαπραγματεύεται με τα άλλα μέρη. Ε, το κοιτάζουμε αυτό ε, συστηματικά. Το είδαμε πρόσφατα στις διαπραγματεύσεις από τον Καναδά. Τώρα σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις μας. Κάποιοι το ε, ανέφεραν και νομίζω ότι εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε θετικά. Ο Επίτροπος Δεχού θα αναλύσει τα αποτελέσματα των σχετικών διαβουλεύσεων στο προσεχές μέλλον. Μα είπατε ότι πρέπει να προσέξουμε πώ θα διαπραγματευόμαστε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τι διαπραγματεύσει αυτέ και ότι πρέπει παρόλα αυτά οι πολίτε και τα ευρωπαϊκά εθνικά κοινοβούλια να τηρούνται ενήμεροι για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και συνομιλιών μα. Για ένα θέμα που ακούστηκε επανειλημμένω, ιδίω από του Έλληνε βουλευτέ. Και το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι ανησυχούν για τα τη Τρόικα. Ξέρετε πώ δημιουργήθηκε η Τρόικα, ξέρετε ότι ήταν ένα εργαλείο για να διαχειριστούμε την κρίση και ξέρουμε, ξέρουμε και ότι ο προπολογισμός της βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε πόσα χρήματα χρειάστηκαν για τα διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό για το οποίο λυπάμαι είναι που σε ό,τι αφορά, για το, πολιτικό, το πολιτικό τίμημα κάθε φορά κατηγορείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Δεν το βρίσκω δίκαιο αυτό. Διότι η κατάσταση πολλών χωρών, ιδίω τη Ελλάδα, δεν ήταν στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλαμε να είναι πολύ καλύτερη. Αγωνιστήκαμε για την Ελλάδα από την αρχή ω το τέλο. Δυστυχώ αυτό δεν αναγνωρίζεται πάντοτε. Επίση, να σα πω ότι επισκέφθηκα την Ελλάδα αρκετέ φορέ του τελευταίου μήνε. Και πιέσαμε όχι μόνο εμεί μάλλον εντυπωσιαστήκαμε όχι μόνο εμεί, όλοι όσοι συμμετείχαν στην ομάδα, από τι τεράστιε προσπάθειε που έχουν καταβληθεί, από τον πόνο που χρειάστηκε να γνωρίσουν οι Έλληνε πολίτε και βλέπουμε ότι επιτέλου έχει περάσει σε θετική ισορροπία η Ελλάδα. Βλέπουμε η Ιρλανδία να ξεπερνά τα προβλήματά τη, βλέπουμε η Ισπανία, βλέπουμε η Πορτογαλία να τα πηγαίνει πολύ καλύτερα με τι εξαγωγέ από ότι εδώ και πολλά χρόνια στην ιστορία. Οπότε να πω απλώς ότι επιτέλους νομίζω οδεύουμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η θετική τάση και ότι οι πολίτες θα το αναγνωρίσουν αυτό. Σε ό,τι αφορά το σχιστολιστικό αέριο, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι έχετε ειδικέ γνώσει για αυτή την κατάσταση θα έχετε σημειώσει ότι είχαμε συστάσει για το σχιστολιστικό αέριο και αυτό ήταν μέρο των μέτρων για την ενεργειακή μα πολιτική που εγκρίθηκε πριν από λίγε εβδομάδε. Είπαμε σαφώ ότι τα ελάχιστα κριτήρια προστασία του περιβάλλοντο θα ισχύουν και ότι σε αυτή τη φάση θα παρακολουθούμε τη διαδικασία πολύ στενά και σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της επικουρικότητας. Τώρα, τα κάτι μελη θα αποφασίζουν εάν θέλουν να συνεχίσουν ή όχι, εάν θα προχωρήσουν σε εξόριξη και οι διαδικασίες αυτές διοργανώθηκαν σε σχετικά σύντομο στο χρονικό διάστημα, ώστε να βεβαιωθούμε για το πώς χρησιμοποιούνται σχετικές τεχνικές και τι περιβαλλοντικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν να ολοκληρώσω λέγοντας κάτι για το οποίο κατά πόσο φαινόταν πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι. Νομίζω ότι πολλοί από εσά το καταστήσατε σαφέ. Θέλω και εγώ να το υπογραμμίσω. Να είμαστε σαφεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη αυτή καθεαυτή, είναι πρωταγωνίστρια στην προστασία του περιβάλλοντο. Θα έπρεπε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχουμε τα πλέον απαιτητικά περιβαλλοντικά κριτήρια παγκοσμίω. Αυτό χάρη στη δική σα τη δουλειά. Στο έργο του Ευρωκοινοβουλίου χάρη στην επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά τι περιβαλλοντικέ μα πολιτικέ, είναι πολύ συγκεκριμένε οι απαιτήσει του Κοινοβουλίου. Ε, το ίδιο και στι περιβαλλοντικέ ε, προτεραιότητε. Θα πρέπει λοιπόν γι' αυτό να καμαρώνουμε. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μπορεί να πει ότι σκοπεύει να παραμείνει ένα παγκόσμιο πρωταγωνιστή λόγω τη υψηλή ποιότητα τη περιβαλλοντική μα πολιτική και στο μέλλον θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας τις ερχόμενες εβδομάδες και τους ε, ερχόμενους μήνες. Ειδικά σε ένα τομέα που συχνά ε, ε, αγωνιζόμαστε ώστε να επανεθνικοποιήσουμε κάποιες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, να ξαναπάμε κάποιες φορές προς τα πίσω ίσως στην ιστορία. Αλλά είναι σημαντικό, είναι σημαντικό σε τέτοιους σοβαρούς Τομεί σε μια τόσο μικρή ήπειρο όπω η Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή λοιπόν κλίμακα, να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις. Και αυτό θα συζητηθεί πιστεύω εκτενώς στην περίοδο της προεκλογική εκστρατεία. Ευχαριστώ πολύ. Ich möchte mich... Θα ήθελα κλείνοντα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της πρώτης επιτυχούς πρωτοβουλίας των πολιτών. Να ευχαριστήσω την κυρία Περέτ η οποία είναι πρόεδρος ε, της ε, πρωτοβουλίας αυτής και τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε καν η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία με τόσο ευρία πρόσβαση και για συμμετοχή και υπογραφή μέσω διαδικτύου, το οποίο το υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχω ε, μια μεγάλη έκκληση και αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό της πρόσβασης στην υδροδότηση και της αποχέτευσης και σε ό,τι αφορά την διάσταση των διαπραγματεύσεων ελευθερίου εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, θα πρέπει αυτό να το έχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού της. Έχουμε ήδη συμφωνίες και σε διάφορες περιπτώσεις το Κοινοβούλιο έχει φροντίσει και έχει εμ, φροντίσει να αποτύχουν πρωτοβουλίες και τέτοιες συμφωνίες. Το νερό και σε ό,τι αφορά τη σχέση του με τον καταναλωτή είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί διαφορετική πολιτική. Θα ενημερώσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σημερινή ακρόαση και για τη στοχοθέτηση. Για όσα συζητήθηκαν εδώ σήμερα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες ε, εξ αριστερών και εκ δεξιών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, σήμερα όμως παραπέθησαν και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα ήθελα στην επόμενη περίσταση να συμμετέχουν εδώ στο πάνελ και εκπρόσωποι ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γιατί ασκήθηκε ε, κριτική στον κύριο Σεύκοβιτς. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να συμμετέχει και το Συμβούλιο προκειμένου και τα τρία όργανα να μπορέσουν να λογοδοτούν, να απαντούν σε ερωτήσεις. Αυτό εγώ θεωρώ άμεση δημοκρατία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα ήταν η πρώτη τέτοια επιτυχής ε, πρωτοβουλία. Να σας διαβεβαιώσω δε, εσάς ως οργανωτές, ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθήσει πολύ στενά το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή την πρώτη πρωτοβουλία, γιατί έχουμε και εμείς το δικαίωμα ε, εκθέσεων πρωτοβουλίας με συγκεκριμένες επιπτώσεις, με συγκεκριμένο αντίκτυπο. Σε περίπτωση ανάγκης λοιπόν θα το ζητήσουμε αυτό. Νομοθετική έκθεση και νομίζω ότι 1,9 ψήφι, εκατομμύρια ψήφι, 1,9 εκατομμύρια ψήφι είναι κάτι το οποίο μιλάει από μόνο του. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Πάρτε το αυτό μαζί σας σαν μήνυμα και ζήτησα να με ενημερώσουν πριν από λίγο η κυρία η οποία ασθένησε, είναι καλύτερα. Ήταν πραγματικά σοκαριστική εκείνη η στιγμή, αλλά χαίρομαι που τα πάει καλύτερα. Να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν και σας παρακαλώ να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη τα οποία ακούσατε σήμερα. Σας εύχομαι καλή επιστροφή στην πατρίδα σας και σας ευχαριστώ πολύ.